Uh, Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Επιτροπής τώρα. Σήμερα έχουμε επαρκή χρόνο να συζητήσουμε ορισμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και έχουμε και τον Επίτροπο Ανάπτυξης, ο οποίος θα έρθει αργότερα για να μας κάνει μια παρουσίαση και να απαντήσει οι ερωτήσεις μας το 16 σήμερα στην ημερήσια διάταξη είναι συστήματα υγείας στην υποσαχάρη Αφρική και η παγκόσμια υγεία. Θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων και μία εξέσταση του σχεδίου εκθέσεως της συγγητρίας και ε, η ημερομηνία για την κατάθεση των τρομολογιών είναι μέχρι 14 Αυγούστου το μεσημέρι η κυρία Βερονίκ Ντεκάιζερ, με συγχωρείτε, 14 Ιουλίου, αύριο, αύριο. Η κυρία Ντεκάιζερ έχει καθοριστεί ως εισηγήτρια σχετικά με τα συστήματα υγείας στην υποσαχάρη Αφρική. Ε, και ε, πρόκειται, έχει ετοιμάσει ένα κείμενο επί του οποίου θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που σας ζήτησα να διορθώσετε την ημερομηνία, αλλά ήταν μια ουσιαστική λεπτομέρεια, διότι μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες και η ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή μας θα γίνει 30 Αυγούστου, την πρώτη μέρα που θα ξαναξεκινήσουμε μετά τις διακοπές. Είναι λοιπόν δύσκολο να γίνει μια συνενετική κοινοβουλευτική δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Και ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση για την έκθεση, η πρώτη μάλλον συζήτηση, έγινε στην τελευταία ολομέλεια του Στρασβούργου. Νομίζω στο Στρασβούργο δεν το συζητήσαμε. Τέλος πάντων. Μία πρώτη συζήτηση έχει γίνει για την έκθεση αλλά το γραπτό κείμενο για λόγους μετάφρασης δεν ήταν διαθέσιμο ακόμη οπότε ανέλαβα τότε την πρωτοβουλία να συναντήσω τους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων με τη σκέψη ότι αν μπορούμε να προχωρήσουμε την ε, εξέταση της εκθέσεως και τις ε, πρώτες ε, διαπραγματεύσεις αφήνοντας τον καθένα την ελευθερία κίνησης θα ήταν καλό. Ε, άφησα λοιπόν σε όλους ο χρόνο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου να συζητήσουμε και προετάθησαν μια σειρά από τροπολογίες λαμβάνοντας υπόψη ότι αύριο θα τελειώσει η προθεσμία. Έχετε δηλαδή ακόμη κάποιο χρόνο και ο καθένας θα έχει χρόνο να διατυπώσει τις απαντήσεις του. Σας υπενθυμίζω το στόχους αυτής της έκθεσης και πρέπει να σας πω ότι ο στόχος μου δεν είναι ε, να κατακρίνω την εξαιρετική δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο ή να συνενέσουμε σε ολόκληρη την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία ε, γνωρίζουμε θαυμάσια αλλά να τονίσουμε απλώς στο θέμα αλληλεγγύης, σε θέματα υγείας, το οποίο σήμερα όχι μόνο ισχύει στην Αφρική με το όνομα του Τονκίν, αλλά έχουν βελτιωθεί, ε, εκλεπτιστεί, υπάρχουν εκατοντάδες ε, τέτοιες μονάδες στην Αφρική με την στήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων ή ασφαλιστικών εταιριών διεθνών. Υπάρχει λοιπόν το σύστημα αλληλεγγύης το οποίο ίσως δεν είναι συνεκτικές. Υπάρχουν, ε, υπάρχει πληθώρα συστημάτων αλλά ο στόχος ήταν να πούνε στην Επιτροπή ότι είναι ένα βασικό σύστημα αλληλεγγύης το οποίο ε, είναι ριζωμένο στην Αφρική και όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή με διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτή είναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο τονίζεται. Το δεύτερο είναι ότι τα συστήματα αυτά των αντασφαλίσεων ή ασφαλίσεων, αμοιβαίων ε, κεφαλαίων, δεν μπορούν ε, να είναι αυτάρκοι από πλευράς χρηματοδοτήσεως και άρα χρειάζεται ε, να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω. Η χρηματοδότηση αυτή πιστεύουμε ότι σύντομα ότι δεν ε, ε, δεν θα μπορέσει σύντομα να καλυφθεί από τις αφρικανικές χώρες σε θέματα υγείας. Γι' αυτό, ε, εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνέχεια και για να μπορέσουν να τους ενθαρρύνουν να καλύψουν στο μέλλον τις δαπάνες τις υγειονομικές και ή να τις στηρίξουμε. Εκεί παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα περαιτέρω ένα πρόβλημα, ίσως δεν είναι πρόβλημα, είναι ένας εμπλουτισμός, ο οποίος όμως μπορεί να καταστεί προβληματικός. Διότι αν δούμε τα κάθετα ταμεία, δηλαδή τα ταμεία τα οποία καλύπτουν ορισμένες παθολογίες που έχουν μεγάλη απήχηση ε, στο δημόσιο χώρο αν μιλάμε για τη ε, φυματίωση, για το AIDS και άλλα αυτά ε, τα θέματα προσελκύουν σημαντικές ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις βέβαια γιατί καταπολεμώντας την ελνοσία παραδείγματος χάνει σώνει κανείς πάρα πολύ παιδιά αλλά έτσι μένουν ελάχιστα χρήματα για άλλες ε, υπηρεσίες βασικές, ε, για αμοιβές αντιμετωπίσεις ε, όπου χρειάζεται μία διαγώνιος ε, αντιμετώπιση. Χρειάζονται ναι μεν οι, τα κάθετα ταμεία αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε τις βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Γι' αυτό και εμείς βασιζόμαστε εις ε, τα θέματα αμοιβαίας στηρίξεως και στα βασικά στοιχήματα. Τώρα, αυτά πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένα, όχι υποχρεωτικά. Διότι σε ορισμένες πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει ενδέχεται να υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Οι βασικές υπηρεσίες είναι οι οριζόντιες, οι συνολικές είναι κάθετες και υπάρχει και μία διεγόνιος η οποία θα ε, επέτρεπε μαζί με τις συνδρομίες των ασφαλισμένων να οδηγήσει στη συγκέντρωση των, ε, της χρηματοδοτήσεως των βασικών υπηρεσιών. Να ε, λεχθεί δηλαδή ορίστε αυτό θέλουμε να κάνουμε, έτσι θέλουμε να συμμετάσχουμε εις τη χρηματοδότηση της υγείας μας, τα κράτη κάνουν ορισμένες προσπάθειες προσπάθειες αλλά και εμείς θέλουμε να εμπλακούμε ή στη χρηματοδότηση των υγειονομικών υπηρεσιών. Οπότε υπάρχει όπως σας είπα η κάθετος και η βασική αντιμετώπιση και αυτή η διαγώνια η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την Αφρική και ε, που συναντούμε και σε πολλές άλλες χώρες. Κάτι δηλαδή δημιουργείται, ε, φυτρώνει, είναι ενδιαφέρον, πρέπει να αναπτυχθεί και σε αυτό βαφισίζεται η έκθεση. Καθότι η ορολογία την οποία να αναφέρω δεν είναι πάντοτε εύκολη γιατί μεταξύ ε, των γαλλοφώνων πρώην γαλλικών απικιών και των αγγλοφώνων χωρών δεν χρησιμοποιούμε τους είδους ε, όρους, δηλαδή ε, στην ε, Γαλλία μιλάμε για αμοιβέ ασφαλίσεις mutuelle d'assurance, ενώ στην Αγγλία μιλάμε για μικροχρηματοδότηση, μικροασφάλιση. Ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε ένα ή δύο όρους και αυτή είναι η εργασία η οποία έχει γίνει μέχρι τούδε. Πιστεύω λοιπόν ότι η αλληλεγγύη, η μη κερδοσκοπική μορφή ε, αυτών των ε, αμοιβαίων ασφαλίσεων δεν πρέπει να προκαλέσει αντιρρήσεις και αντιθέσεις ή στην Επιτροπή μας. Υπάρχουν βέβαια τα θέματα που έθιξα με τους σκιώδεις και που ξέρω ότι είναι ευαίσθητα. Η βοήθεια την οποία ε, εμείς ε, συζητήσαμε διότι θεωρήσαμε ότι για αυτές τις αμοιβέ ασφαλίσεις οι ε, οριζόντιες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτουν την αναπαραγωγική υγεία και πιστεύω ότι η καταπολέμηση του AIDS, η δυνατότητα για τις Αφρικανές να επιλέξουν μόνες τους τη στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο θα, δώσουν, θα φέρουν στη ζωή τα παιδιά τους, τα αντισυλληπτικά, τα προφυλακτικά, είναι ε, οι διαμάχες, η υψηλή παθολογία του AIDS, AIDS, το θέμα της αναπαραγωγικής υγείας που δεν είναι ε, θέμα ιδεολογίας αλλά θέμα της ε, προστασίας της ζωής. Υπάρχει μια τεράστια θνησιμότης, μεγάλη παθολογία για το AIDS και πιστεύω ότι εδώ μιλάμε για ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα το οποίο προσπαθώ να τονίσω για ορισμένους συναδέλφους οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις ε, στο θέμα αυτό και συμφωνώ μαζί τους ε, και σέβομαι μεν τις απόψεις τους αλλά δεν συμφωνώ. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις τροπολογίες εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία. Ορισμένα οι τροπολογίες αναφέρονται εις ε, τα ε, βασικά θέματα που έθιξα δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές ε, συμβιβαστικές λύσεις αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να τροποποιήσω την έκθεσή μου εάν μου το ζητήσετε. Ευχαριστώ κυρία Ντεκάιζερ. Προφανώς έχετε κάνει εξαιρετική εργασία και θα έπρεπε να σας πω ότι ο Επίτροπος θα έρθει στις 4. Έχουμε δηλαδή 40 ε, λεπτά για να συζητήσουμε την έκθεσή σας. Και θα προσπαθήσω να το τραβήξουμε όσο μπορούμε πιο μακριά. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Κάσμα να αρχίσει με τη γενικότερη συζήτηση. Για να σας βοηθήσω, αντί να συνεισφέρω στη συζήτηση, Ίσως θα πρέπει να αρχίσω διαβάζοντας την καταιγίδα του Σέιξπιρ και να προχωρήσω στο, στα συμπεράσματα, αν δεν θέλετε να διακόψουμε για καφέ. Είναι ε, ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η έκθεση. Ε, προτρέπει τη Βελγική Προεδρία να συζητήσει το όλο θέμα, αν όχι στις Επιτροπές, τουλάχιστον στην Ολομέλεια. Και θα ήθελα Μιλώντας ήδη στη Βερονίκ, θα ήθελα να προβάλλω μία τροπολογία μίας μόνο γραμμής για να μιλήσουμε για το καθολικό παγκόσμιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όπως υπάρχει στη Σουηδία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία έτσι ώστε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στα διάφορα μοντέλα, στα διάφορα πρότυπα να μην προβάλλουμε το ένα ή το άλλο, διότι όλα επηρεάζουν, το καθένα με τον τρόπο του. Γι' αυτό υπάρχουν επιλογές. Θα ήθελα να υποβάλω μία τροπολογία, μία πολύ απλή. Μεταξύ των παραγράφων 16 με 18. Δυστυχώς αυτά έχω να σας πω αφού δεν θέλετε την καταιγίδα του Σέξπιρ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα πρέπει, αν θέλετε να καλύψουμε χρόνο, μπορούμε να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο που οδήγησε στη δόξα της Ισπανίας και οδήγησε σε μια αισιοδοξία που είναι πολύ ε, χρήσιμη για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στη Νότια Αφρική, από την Νότια Αφρική μέχρι την Ισπανία. Θα ήθελα όχι να καλύψω το χρόνο, αλλά να μιλήσω για τη σημασία αυτής της έκθεσης και να δούμε ποιο είναι το υπόβαθρο των προθέσεων της Βερονίκ και όσων ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό. Άρα, το υπόβαθρο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε καινοτόμο, ένα καινοτόμο μέλλον και μια κινητικότητα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τις καταστάσεις έλλειψης ανάπτυξης. Δεν αρκούν τα μεγάλα κριτήρια και οι μεγαλεπίβολες ε, εισφορές του προϋπολογισμού αλλά θα πρέπει να βρούμε και νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω συστημάτων φορολόγησης και εισφορών και να βρούμε και να εξεύρουμε και νέους τρόπους διαχείρισης με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών, των συνεργειών και του τρόπου που έχουν οι κοινωνίες ε, να αντιμετωπίσουν τα επιμερούς θέματα. Θα ήθελα να πω προς τον κύριο Ντέβα ότι ένας μεγάλος ε, θεωρητικός ε, Άγγλος, ο Βίργο Πάρεκ, ο οποίος ζει στην Ινδία, είπε ότι δεν υπάρχει μεμονωμένη λύση των προβλημάτων, διότι υπάρχουν διαρθρώσεις οικογενειακές, πολιτικές, οι οποίες είναι πιο συλλογικές και εστιάζουν την προσοχή σε περισσότερα επιμέρους θέματα μεταξύ συντονισμού, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Άρα δεν μιλάμε για μεμονωμένη και μοναδική επίλυση προβλημάτων. Γι' αυτό συμφωνώ με τη Βερονίκ ότι θα πρέπει να βρούμε μια συλλογική αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και υγιεινής, δηλαδή να έχουμε ένα συλλογικό σχήμα αλληλεγγύης, ιδιαίτερα εκεί που το κράτος έχει αποτύχει, η κοινωνία έχει αποτύχει και θα πρέπει να βρούμε αυτή τη μεγάλη διαγώνιο η οποία διατρέχει όλα αυτά τα συστήματα μεταξύ ενός ε, ε, γενικευμένου συστήματος υγείας, τα οποία, το οποίο είναι ασθενές, ή εγκάρσια συστήματα διαχείρισης που οδηγούν από πάνω προς τα κάτω, παρά οριζόντιες ε, επιλύσεις. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε όπως εξέφρασε και η Βερονίκ. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα υποβάλω μία τροπολογία, αλλά περισσότερο από τροπολογία είναι μία σκέψη που θα πρέπει να διέπει το σύνολο των θεσμικών οργάνων και την Επιτροπή μας. Δηλαδή, όταν υπάρχουν πόροι στα εγκάρσια ταμεία και όταν μιλάμε για συγκεκριμένες αδυναμίες συγκεκριμένων χωρών, τη στιγμή που προβάλλεται η επίλυση του προβλήματος και έρεται η αδυναμία, θα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές σωτηρίας με βάση αυτά τα εγκάρσια ταμεία για να μπορούμε να κινηθούμε σε άλλες χώρες ή άλλες αδυναμίες που να έχουν επίσης κάθετο εγκάρσιο χαρακτήρα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ήθελα μόνο να καλύψω χρόνο, αλλά ήθελα να τονίσω και να υποστηρίξω αυτή την προοπτική. Όχι καινοτόμο πάντα, διότι υπάρχει σε πολλές περιφέρειες της Αφρικής, αλλά να ενισχύσω αυτή την προοπτική συλλογικής επίλυσης των προβλημάτων υγείας, στις χώρες όπου τα εθνικά συστήματα είναι αδύναμα συστήματα, διότι τα κράτη είναι αδύναμα και η κεντρική κυβέρνηση είναι αδύναμη. Νομίζω λοιπόν ότι η υγεία είναι ένα στοιχείο, είναι μια βασική συνιστόσα, μια βασική φυσική συνιστόσα, η οποία όμως φέρει και ένα ψυχολογικό τμήμα και αυτή η έννοια της αλληλεγγύης, η συλλογική αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί, πέρα από την ιατρική περίθαλψη, πέρα από τις τεχνολογίες, είναι ένας ιδιαίτερα σημαίνων παράγων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες αυτές. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνεισφορά Θα ήθελα ο Τσαρλ Κόρενς τώρα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα, ο Επίτροπος που θα καταφτάσει, θα στις 4, οπότε ε, καλό είναι να συνεχιστεί η συζήτηση μέχρι τότε. Δεν είμαστε και πολλοί εδώ για να αγωνιζόμαστε για να πάρουμε το λόγο, οπότε ας λίγο τη συζήτηση για να περάσει ο χρόνος. Ε, γιατί εγώ τα έχω πει με την κυρία Ντεκέιζερ στο Στρασβούργο ήδη. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν γιατί θα επαναλάβω αυτά που είπα. Είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση, εξαιρετικά επίκαιρη. Είναι ένα φυτόριο ιδεών και καλό είναι να διερευνήσουμε αυτές τις ιδέες τα επόμενα χρόνια. Εφόσον λοιπόν προτίθεμαι να διευρύνω τη συζήτηση, αρχίζοντας ε, θα συγχαρώ τον συνάδελφο Γκερέιρο για το παγκόσμιο κύπελο που κερδίσανε ε, την ε, Κυριακή. Για να επανσυνδέσω ότι το παγκόσμιο κύπελο με το θέμα μας, θα έλεγα ότι όλοι προπονούνται και κινητοποιούνται με τα παγκόσμια κύπελα. Κοιτάξτε τι έγινε στην Νότια Αφρική τις τελευταίες πέντε εβδομάδες ε, προέβαλε μια διαφορετική εικόνα η Αφρική σε σχέση με αυτή που έχουμε συνήθως ε, για την Αφρική που όλα γίνονται στο πόδι. Ε, υπήρξα, υπήρξε λαϊκή κινητοποίηση, όλοι ήταν μπροστά στις γιγαντοθόνες που βρίσκονταν σε στρατηγικά σημεία Υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός από τα εκατομμύρια τηλεθεατών και επισκεπτών. Με τις βουβουζέλες λοιπόν, με αυτό τον εκοφαντικό ήχο, εμψυχώσαμε όλοι το κύπελο. Καλό είναι λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου τη μεταφορά μπορούμε να κάνουμε και την παρομοίωση με τον παγκόσμιο κύπελο. Υπήρξαν καταπληκτικές επιδόσεις τις τελευταίες εβδομάδες ε, Κανείς δεν είχε ποντάρει στην ικανότητα να ε, καταλήξουμε σε συνθήκες ασφαλείας που επιθυμούσαμε. Κανείς ε, δεν είχε μαντέψει ε, ότι η Νότια Αφρική θα τα κατάφερνε να οργανώσει με αυτόν τον τρόπο το παγκόσμιο κύπελο. Ανακαλύπτουμε ξαφνικά μία νέα Αφρική. Μέχρι στιγμής τη σκεφτόμασταν το AIDS, της διάφορες ενώσους, το AIDS, της συγκρούσεις ανάμεσα στις ε, αφρικανικές φυλές, ε, στις διάφορες εθνότητες. Και τώρα όμως άλλαξε η εικόνα της Αφρικής. Ε. Μπορεί η Αφρική, το απέδειξε, να αναλάβει μια καταπληκτική διοργάνωση. Από την περασμένη Κυριακή μετά έχει κατοχυρωθεί αυτή η νέα εικόνα της Αφρικής. Αν ο κύριος Πίμπαλξ ερχόταν στις 4.30 θα σας έκανα και ένα λογίδριο για την ενότητα της Ισπανίας. Ε, τώρα πραγματικά έχετε, είσαστε όλοι Ισπανοί ενωμένοι όπως ποτέ στο παρελθόν. Προτείνω λοιπόν στο Βέλγιο, στο μέλλον, ε, να ε, συμμετάσχει με μεγαλύτερη ζέση, με μεγαλύτερο ζήλο σε όλους τους διαγωνισμούς. Ε, θα ήταν να κερδίσουμε και το πρωτάθλημα. Η Αφρική τόλμησε λοιπόν. Η Αφρική ακολούθησε νέους δρόμους. Δεν ακολούθησε την πεπατημένη. Αυτό είναι το βασικό δίδαγμα του κυπέλου. Όλα τα προβλήματα ε, με κάποιο τρόπο συνδέονται με την Αφρικανική Ήπειρο ε, και κυρία Ντεκέιζερ, ε, η έκθεσή σας με βρίσκει απολύτως σύμφωνο σε όλα τα σημεία. Θα ήθελα λοιπόν να αναπτύξω κάποια επιμέρους σημεία. Η κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή την προσέγγιση των συνεταιρικών οργανώσεων. Στο Χονγκ οι εκπρόσωποι του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας ε, είπαν ότι δεν αναπτύσσεται το εμπόριο στην Αφρική επαρκώς για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι για να εξυπηρετηθούν οι ευρωπαϊκές αγορές ε, πρέπει να διατεθεί ένα φάσμα προϊόντων που ενδέχεται να καταναλωθούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Στη ΣΥΠΑ, παραδείγματο χάρη, αλλάζουν τα γούστα των καταναλωτών συχνά και άρα τι πρέπει να γίνει η προσαρμογή της παραγωγής σε αυτήν την εξελεκτική διαδικασία για να ικανοποιεί το καταναλωτής. Αλλά πρέπει κάποιος να διακινδυνεύσει για να φέρει τις αλλαγές αλλά σκέφτονται όλοι τον κίνδυνο και δεν ρηψοκινδυνεύουν. Το ίδιο συμβαίνει και με την κοινωνική ασφάλιση. Αυτοί που νοσούν, αυτοί που έχουν πάθει ατύχημα, που πάσχουν από κάποια αναπηρία, πρέπει να βοηθηθούν, αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα από οικονομική πλευρά και μόνο. Πρέπει να προαγάγουμε αυτά τα ε, συστήματα ε, υγειονομική ε, περίθαλψης προτείνοντα την έκθεσή σα. Δεύτερον, όπως έχω πει, ε, οφείλουμε να τονίσουμε την περιφερειακή προσέγγιση. Όπως και στην Αφρική και όχι μόνο στην Αφρική, α αρχίσουμε από τις δικές μας χώρες. Πρέπει να γίνει η καταγραφή της προσφοράς, της ζήτησης και να δούμε αν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο. Στην Αφρική βέβαια δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι εδώ ακόμη ο κύριος Επίμπαλξ, οπότε μπορεί να επαναλάβω και κάποια σημεία ε, που έχω ήδη αναφέρει. Ε, στο Νίγηρα, παραδείγματος χάρη, άμα έχετε μια, ένα μευτήριο ε, και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Νιγηρίας, αν έχετε άλλο με ευτήριο που κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, προσφέρει ακριβώς οι ίδιες υπηρεσίες, υπάρχει απώλεια πόρων. Δεν χρειάζονται και τα δύο. Θα πρέπει να είναι αλληλοσυμπληρούμενοι οι πόροι ε, της Αφρικής. Και εφόσον αυτά ε, τα δύο νοσοκομεία είναι σε δύο διαφορετικές χώρες, ακολουθούνται δύο διαφορετικές ε, πολιτικές στον τομέα της υγείας. Οπότε χρειάζεται διάλογος ανάμεσα στι γειτονικέ χώρες, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να είναι αλληλοσυμπληρούμενοι πόροι. Χρειάζεται λοιπόν μια χαρτογράφηση υγειονομική, α το πούμε έτσι, που θα καλύπτει όλη την ε, περιοχή. Κάτι άλλο μπορεί να φαίνεται ε, χωρίς σημασία, αλλά έχει βαρύτητα. Στο Μπούρκινα Φαζό και στο Μαλί, παραδείγματο χάρη, επιδιώκουν να έχουν κοινό σύστημα ε, για τα ασθενοφόρα. Πολύ καλό παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας για τη διακομιδή των ασθενών. Ε, άλλο παράδειγμα που καταδεικνύει ότι πρέπει να υπερβούμε την εθνική αντιμετώπιση. Το θέμα των ιατρών. Σε κάποιε χώρε υπάρχουν ε, δομέ στον τομέα τη υγεία, υποδομέ, αλλά δεν υπάρχουν ε, αρκετοί γιατροί. Μα είναι παράλογο. Στη Ρουάντα, παραδείγματο χάρη, στη Γουαμαγκανά, υπάρχει υποδομή, υπάρχει νοσηλευτική μονάδα, αλλά κανένα γιατρό. Ε, και θέλαν, θέλαν να προτείνουν, ε, να προαγάγουν μια θεραπεία για τους ε, ασθενείς του AIDS. Ναι, όλα αυτά καλά, αλλά δεν υπήρχαν γιατροί για να χορηγήσουν τις θεραπευτικές αγωγές, τις αντιρετροϊκές αγωγές. Χρειάζονται σημαντικοί πόροι. Κινητοποιήθηκε βέβαια το Υπουργείο Υγείας ε, στη Ρουάντα για να ε, ε, βρεθεί ένας γιατρός, μετά απευθύνθηκαν στους ομογενείς στη Διασπορά και στην Αφρικα... κοινότητα Αφρικανικών κρατών στη συνέχεια για να βρεθούν γιατροί. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί λοιπόν. γιατί δεν είναι επαρκή οι αποδοχές τους. Ε, οπότε, εάν Το καλό θα ήταν ε, να ε, μετεκπαιδεύονται στην Ευρώπη και να επιστρέφουν στη χώρα τους ε, και να κάνουν τακτικά ταξίδια αν υπάρξει ένα είδος συνεργασίας, ένα είδος εταιρική σχέση ανάμεσα στην χώρα καταγωγής και κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο ένα πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι σχολίασα ήδη τα τρία κατά με βασικά σημεία της έκθεσης, οι γιατροί, η περιφερειακή διάσταση και η εμπειρία. Θέλω να ζητήσω να ρωτήσω κάτι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα ήταν άνισο να περιμένετε από εμά να γεμίσουμε το χρόνο μέχρι τις 4 Οπότε, κυρία Ντεκέιζερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Μήπω θα έπρεπε να κινήσουμε μια πιλωτική διαδικασία από κοινού με τον, ε, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για να κάνουμε μια αξιολόγηση ε, για αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει, κυρίως ε, για, ε, υπόψη αυτή την περιφερειακή διάσταση που προανέφερα. Ε, γιατί αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να πραγματευτεί το ζήτημα υπό την περιφερειακή διάσταση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να χρησιμοποιηθούν εταιρικέ σχέσεις με μια νότια χώρα και εμείς μπορούμε να συνοδεύσουμε την όλη διαδικασία, να την παρακολουθήσουμε από κοντά. Ζητώ συγγνώμη που δεν μίλησα παραπάνω, ήμουν υπερβολικά σύντομος, αλλά ελπίζω να κατάφερα να συμβάλλω ούτως ώστε να κρατήσει η συζήτηση μέχρι τις 4. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα σοφά ε, λόγια από έναν πρώην Υπουργό Ανάπτυξης του Λουξεμβούργου. Μετά από τα επενετικά σας λόγια ποτέ δεν θα σας επιπλήξω ή δεν θα μιλήσω άσχημα για σας. on one occasion Θυμάμαι όταν ήμουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ήρθε σε μένα ο WIP που μου είπε ότι πρέπει να ε, έρθεις να κάνεις μία ομιλία γιατί προβλεπόταν στις 10 αλλά θα γίνει ε, στις 7. Θα Πρέπει να μιλήσει για τρεις ώρες για τους μισθούς των δικαστικών. Και του είπα, δεν ξέρω τίποτα για τους μισθούς των δικαστικών. Τώρα, τη στιγμή που έχουμε άλλους συναδέλφους όπως η κυρία Ζαβόσκα και θέλουμε και να ακούσουμε και από τον Επίτροπο, θα ήθελα και εγώ να κάνω ένα σχόλιο προς ε, την εισηγήτρη. Ξέρετε ότι προέρχομαι από τη Σρι Λάνκα, εκεί γεννήθηκα. Και αν δείτε το δίκτυ θνησιμότητας, το προσδόκιμο ζωής για μια γυναίκα είναι τα, 20, τα 82 χρόνια, ενώ για του άντρε είναι 78, στη Σρι Λάνκα όλα αυτά. Αλλά αν δείτε τους ίδιους δείκτες το 48 ε, κατά την ανεξαρτησία ήταν 56 και 64 αντιστοίχως. Άρα έγινε κάτι τα τελευταία 60 χρόνια για να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στα δυτικά πρότυπα. Και το ένα που έγινε ήταν η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο ε, έδινε δωρεάν, παρήχε δωρεάν υπηρεσίες και προληπτικά και προληπτικές ε, υπηρεσίες, μάλλον υπηρεσίες πρόληψης έτσι ώστε μέσα στη ε, διαδικασία πρόληψης να αποφεύγονται ασθένειες και να μην θεραπεύονται. Και η παιδική θνησιμότητα έπεσε και έφτασε τα δυτικά πρότυπα. Άρα ήδη κατά την εγκυμοσύνη οι γυναίκες κάνουν προληπτικούς ελέγχους για να δούνε πώς θα αντιμετωπιστεί η οικειοφορία. Αυτό το, θέμα, αυτό το σχέδιο δεν είναι και τόσο ακριβό και ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πείρα ορισμένων κρατών όπως στη Σρι Λάνκα, για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ε, ε, διαφορετικά πρότυπα. Βεβαίως και ο ΠΟΗ έχει ε, διαφορετικές συγκριτικές μελέτες εθνικών συστημάτων υγείας, για να δούμε κατά πόσο η προληπτική υγεία είναι αποδοτική ως προς το συνολικό κόστος και έτσι προλαμβάνονται ασθένειες. Εμείς το κάνουμε τώρα εδώ αυτό σε σχέση με τη χορήγηση ασπιρίνης για την αποφυγή ε, ε, του ενθράγματος ή ε, παρενφερής αντιμετωπίσης ασθενειών. Η κυρία Σαμπόρσκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πραγματικά περίπλοκο θέμα το οποίο ε, πραγματεύεται η έκθεση αυτή και η, η συγγήτρια ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στις υποανάπτυξη χώρες, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι λύσεις. Ε, αυτό που με εκπλήσει είναι η μορφή με την οποία έχει συνταχθεί η έκθεση αυτή και ε, το επικροτώ. Έχω όμως ορισμένα ερωτήματα. Μιλάτε για ένα συνέδριο που έγινε στην Μπουρκίνα Φάσο το 2008 και όπου οι αφρικανικές χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση ότι 15% του προϋπολογισμού τους θα διετίθετο για την υγεία. Είναι ένας υψηλός αριθμός ε, και εδώ μιλάμε για διάφορες ε, χώρες και πρέπει να δούμε πόσο μεγάλο ε, είναι το επίπεδο του κρατικού προϋπολογισμού για να υπολογίσουμε ποιο ποσοστό χρησιμοποιείται. Στο σημείο 5 για την αναπαραγωγική ε, υγεία βλέπω ότι αναφέρεστε στα δικαιώματα των γυναικών και ότι υπάρχει πίεση για να μπορούν να αποφασίσουν μόνος τους για την αναπαραγωγική τους υγεία. Ουσιαστικά ε, βασικό είναι ε, η γυναικολογική περίθαλψη και η βοήθεια κατά τον ε, τοκετό ε, διότι την περισμένη εβδομάδα συζητήσαμε στο Στρασβούργο για το AIDS και είπαμε ότι είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Ξέρουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια διαθέτει πάρα πολλά χρήματα ε, για την έρευνα στον, ε, στον τομέα αυτό. Γιατί λοιπόν είναι τόσο χαμηλός ο αριθμός όλο ο, μιλάμε για μείωση των αριθμών, ακούμε όμως ε, για δισεκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Βερονίξε, τι οφείλεται αυτό. Και έχω μία ερώτηση ε, και σε ένα προλαλήσαντα. Ε, ε, σύμφωνα με την... Μάλλον έχω μία ερώτηση αντίστοιχη με αυτή που έθεσε ένας προλαλήσας. Δηλαδή ε, τι ποσό θα χρειαστεί για να βελτιωθεί η κατάσταση στην Αφρική. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία ζητούν ε, συνδρομή για διάφορες ε, ασθένειες, για ασθένειες που πλήττουν ιδίως τις γυναίκες ε, για τις ε, επιπτώσεις ε, του τοκετού για τους βιασμούς και άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτεί στα τα προγράμματα αυτά διότι δεν ασχολούνται με την αναπαραγωγική υγεία. Δεν αντιλαμβάνουμε πώς τα θέματα αυτά του βιασμού και των τοκετών δεν έχουν σχέση με την αναπαραγωγική υγεία. Θα έπρεπε λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, επιμόρφωση των ε, εντοπίων ε, ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, διότι υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθεί επιμόρφωση γιατρών στην Αφρική. Δεν ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό από την Κούβα και την Κίνα που δραστηριοποιείται στην Αφρική. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, γιατρούς και αυτοί που ασχολούνται με το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στηριχθούν. Σας ευχαριστώ για την έκθεση και προσβλέπω στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ε, τέθηκε ένα σημαντικό ερώτημα. Ε, το περιοδικό Economist πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες ανέφερε ότι 100 ε, εκατομμύρια περισσότερα έμβρια έμβρια κοριτσιών αποβάλλονται από ότι αγοριών. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μέσω των αμβλώσεων θανάτωση πολλών γυναικών διότι εάν το μωρό είναι, είναι κορίτσι και όχι ε, αγόρι ενδέχεται, το έμβριο είναι κορίτσι και όχι αγόρι, ενδέχεται να υπάρξει άμβλωση. Ε, τι γίνεται λοιπόν, διότι αντιλαμβάνουμε ότι ε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη καθόλου σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επανέλθει. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τι ερωτήσει. Δεν θα προσπαθήσω να κερδίσω χρόνο. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση γιατί σχετίζεται με ένα τομέα ε, στον οποίο προσδίδω μεγάλη σημασία. Είναι ένα παλαιό θέμα και η έκθεση αυτή ο οδηγεί στην επικαιροποίηση ενός θέματος που μας ενδιαφέρει. Δεν θα σας μιλήσω για, τα, για το παγκόσμιο κύπελο. Το 87 ήμουνα πολύ άρρωστη και θεωρούσα ότι δεν θα μπορέσω πια να ταξιδέψω και ο πανεπιστημιακός καθηγητής που με παρακολουθούσε και προωθούσε τη συνεργασία με την Αφρική, ήταν μεγάλος ουρολόγος, μου είπε Εάν ε, θεραπευτείτε θα έρθετε μαζί μου στην Αφρική. Και μου είπε ότι τότε θα πρέπει να μοιραστείτε τη ζωή που ζω εγώ. Και πρόκειται για μια ομάδα πανεπιστημιακών γιατρών, εκεί όπου δίδασκα και εγώ. Ήταν εξαιρετική η εργασία τους, και στην ουσία ε, τι έκαναν σε περίπτωση, κατά την περίπτωση το κετού επειδή ε, η γυναίκα μπορεί να... Συρίγγια. Να αποκτήσει Συρινγια ο γιατρός έπρεπε να ε, ράψει στην ουσία αυτά τα σχισίματα που δημιουργούνταν, δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια του το, τοκετού. Τότε δεν υπήρχαν νοσοκόμοι στα διάφορα νοσοκομεία και έτσι στην Αφρική, εκεί που δεν υπήρχε νερό, που δεν υπήρχαν νοσοκόμα για ένα μήνα, βοήθησα σε αυτό το, το ράψιμο μετά την, ε, τον τοκετό και ρωτούσα γιατί οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ε, γεννούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί οι γυναίκες δεν έχουν κέντρα προληπτικής ιατρικής. Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Πρόεδρε. Και ε, επίσης διάφορα αγροτικά ας πούμε κέντρα περίθαλψης και αναρωτήθηκα πώς έχουν δημιουργηθεί τα διάφορα κέντρα υγείας θεωρώντας ότι αυτός ο συγκεντρωτισμός είναι πολύ αρνητικός για, τις, ε, για, τις ε, βασικές, ε, για τη βασική περίθαλψη. Γι' αυτό και το πρωταρχικό σύστημα υγείας αφορά, μάλλον ανέρχεται σε μία τριακονταετία πριν. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Τέβα, ο οποίος μου λέει ότι υπάρχουν ε, γυναίκες που ε, σκοτώνουν το έμβριο γιατί θα γεννηθεί κορίτσι. Αυτό βεβαίως μας, ε, μας αποτροπιάζει, μας οδηγεί σε αποτροπιασμό. Και εκεί που υπάρχει υπέρηχος, πολλές φορές οι άνδρες όταν βλέπουν ότι οι γυναίκες οφορούν ένα κορίτσι και όχι αγόρι θέλουν να το θανατώσουν. Άρα στην Αφρική τουλάχιστον πρέπει κανείς να πάει πολύ μακριά για να βρει ε, υπέρηχο. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει να υπάρχει προληπτική ιατρική και περίθαλψη κατά την κοιοφορία, διότι πολλές ε, γυναίκες ε, θέλουν να κυοφορήσουν κάτω από σωστές συνθήκες. Υπάρχουν δηλαδή όμως συνθήκες όπου οι γυναίκες δεν το επιθυμούν αυτό. Μιλάμε για συνθήκες ε, φτώχειας, μιζέριας, βιασμών και βεβαίως ε, κανείς δεν θέλει να, καμία γυναίκα δεν θέλει να κυοφορήσει όταν έχει υπάρξει θύμα βιασμού κατά τον εσωτερικό εκτοπισμό της και έχει δικαίωμα να αποφασίσει. Κύριε Γκέρενς, Σάρλ, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε ένα δελτίο ιατρικής περίθαλψης και στη συνεργασία μου γνώρισα ολέθριες πρακτικές. Δηλαδή χρηματοδοτούμε τους ε, γιατρούς ε, οι οποίοι ε, προβάλλουν συγκεκριμένα αντίτιμα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας, να μας απασχολήσει το ζήτημα πολύ ε, σοβαρά. Νομίζω ότι η βίζα πολλαπλών εισόδων είναι μια ιδέα την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Δεν θέλω να σας ε, διηγηθώ τη δική μου ζωή αποκλειστικά. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για την χρηματοδότηση των, ε, της βασικής περίθαλψης και τι πόροι θα διατίθενται και ποια είναι τα ε, σενάρια μέσα στα πλαίσια του Global Fund για το AIDS, την ε, φυματίωση και την ελονοσία που θα λάβει η χώρα στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2010. Τι προτίθεται να κάνει, γιατί θα ήθελα να λάβει θέση, η οποία να είναι μια στεναρή θέση. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια χρηματοδότησης των αφρικανικών χωρών. Βασιζόμαστε σε σαφείς δείκτες. Δηλαδή λαμβάνουν υπόψη το, το φόρτο της ασθένειας για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος τους ε, πληθυσμούς, τους ε, πρόωρους θανάτους και ούτω καθεξής και κατά πόσο αυτή η χρηματοδότηση γίνεται με βάση ποσοτικά κριτήρια ή άλλα πολλαπλά κριτήρια. Εντάξει, Εξάντλησα το χρόνο, είναι 4 η ώρα, θα έρθει ο Επίτροπος σε πολύ λίγο. Είναι πολύ ωραίο να έχει κανείς ε, την πολυτέλεια του χρόνου. Πολύ με, πολύ με χαροποίησε αυτό. Χαίρομαι και που ο Ντέβα είναι πρόεδρος, προεδρεύει. Για μια φορά, γιατί περίμενα μεγαλύτερη έφοδο από εκείνον και διαφορετική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση. Ο κύριος Πι ε, περιμένει έξω. Άρα έχουμε τρία λεπτά για να απαντήσουμε. Ο κύριος Σιμένκ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ γιατί δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε γραπτός, εάν το επιθυμείτε θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια ως προς την έκθεση έτσι ώστε να εισαχθούν ορισμένα ε, σχόλια. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και συμφωνούμε στην εστίαση αυτή στα εθνικά συστήματα υγείας, διότι τα συστήματα υγείας έχουν τέσσερις συνιστώσεις το ε, ε, εργατικό δυναμικό, την ε, χρηματοδότηση και τον τρόπο αντιμετώπισης ως προς την πρόληψη και τη θεραπεία. Θα πρέπει λοιπόν ως προς το εργατικό δυναμικό να έχουμε μία κοινότητα για την περίπτωση έλλειψης προσωπικού και θα πρέπει να αναφέρεται αυτό και στο κείμενο για να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις ως προς τις επενδύσεις για την κατάρτιση. Ως προς το εγχώριο προσωπικό, εμείς επενδύουμε αδρά. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους για την επέκταση της αποδοτικότητας έτσι ώστε οι χώρες να ξέρουν ποιο είναι το εμπλεκόμενο κόστος που αφορά την πρόσληψη προσωπικού. Ως προς τη χρηματοδότηση καθεαυτή των συστημάτων υγείας, από όσο γνωρίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες περιφέρειες, δεν υπάρχει ένα σύστημα, ένα ενιαίο σύστημα που να αρμόζει σε όλους και εμείς μαζί με τα κράτη-μέλη επιτελέσαμε ένα μεγάλο μέρος εργασίας. Το παράδειγμα της Σρι Λάνκα είναι πολύ καλό, διότι ξέρουμε από την πείρα μας στην Ασία ότι η κλιμακωτή πρόσβαση σε συστήματα υγείας γίνεται με βάση φορολογούμενα συστήματα, συστημάτων φορολόγησης ή μέσω κοινωνικής ασφάλισης με επιδότηση των φτωχών θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας ευρύτερα και να επικεντρωθούμε στις ε, χρηματοδοτήσεις out of pocket μαζί με την προχρηματοδότηση αλλά θα πρέπει να δούμε την άμεση και την έμεση φορολόγηση όπως ε, εμπλέκεται σε μηχανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Από το 15% από την Αμπούτζα στα εθνικά, επένδυση εθνικά συστήματα υγείας, ξέρουμε ότι υπάρχουν 4 με 5 χώρες που φτάσανε σε αυτό το επίπεδο της χρηματοδότησης, της μερικής κρατικής χρηματοδότησης. Ξέρουμε ότι ως προς τις πληρωμές out of pocket, εντός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας. Και αυτό ίσως είναι μια καλή μνήα που θα πρέπει να γίνει στην ε, έκθεση. Μπορώ να επανέλθω αν θέλετε. Εάν θέλετε μπορώ να επανέλθω γραπτός. Thank you, for uh, Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ντέφα. Τώρα θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον επίτροπό μας, τον κύριο Πίμπαλξ. Uh, it, now great... Με μεγάλη χαρά και το εννοώ, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Θα θυμόσαστε ότι την τελευταία φορά που ήταν εδώ ο Επίτροπος, ένα μήνα πριν, είχαμε ένα διαρθρωμένο διάλογο για τις νομοθετικές εξουσίες το 2011 και ορισμένα μέλη εξέφρασαν τη λύπη τους, διότι δεν μπορούσαμε να προβούμε σε μία ανταλλαγή απόψεων. Όταν λοιπόν είδαμε ότι είχαμε χρόνο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ήρθαμε σε επαφή με τον Επίτροπο και είμαστε ε, ιδιαίτερα ευγνώμονες διότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ε, ήρθατε εδώ για να μας μιλήσετε. Από την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ συνέβησαν πολλά που έχουν μεγάλη σημασία στον τομέα της ανάπτυξης. Θα ήθελα να σχολιάσετε δύο από τα θέματα πριν δώσω το λόγο στους βουλευτές. Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 17ης Ιουνίου όπου συζητήθηκε η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη κορυφής για, την, ε, για τους στόχους της χιλιετίας και την προπαρασκευή της Επιτροπής για τη διάσκεψη το Σεπτέμβριο στα Ηνωμένα Έθνη ως προς τη, τους στόχους ε, της χιλιετίας και ιδιαίτερα πώς αντιμετωπίσατε τις συστάσεις του Κοινοβουλίου ως προς την έκθεση Κάσμαν, προετοιμάζοντας τη διάσκεψη κορυφής. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Πίμπαλξ. Αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε πολύ σημαντικές αποφάσεις επειδή το 2010 είναι ένα πολύ σημαντικό έτος για την ανάπτυξη και τη συνεργασία και ιδιαίτερα για τους στόχους της χιλιετίας. Φοβόμασταν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο γενικότερα θα ήταν κάπως δηλό στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας αλλά τα πιο σημαντικά αποτελέσματα ήταν ότι αναβλήθη, μάλλον αναλύθηκαν και άλλες δεσμεύσεις και επιτελέστηκε πρόοδος και επιτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ετησίως. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα προβάλλουμε αυτή τη βοήθεια, διότι δεν έχει σημασία να ε, προβάλλουμε προτάσεις ε, αργά, γιατί μιλάμε για 0,7% του ΑΕΠ. Και αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν ε, τις πολιτικές τους για μια πραγματική αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης ενέκρινε τις συμπεράσματα του Συμβουλίου με βάση το, το, σχέδιο 12 σημείων, ιδιαίτερα για ευάλωτες χώρες. Uh, για να δούμε πώς εκπληρώνονται οι στόχοι της χιλιετίας, ιδιαίτερα για τα νήπια μέχρι 5 ετών. Άρα ε, συνεισέφερε και η Επιτροπή σας. Ένα πολύ σημαντικό σημείο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ε, στόχων της χιλιετίας. Αυτό είναι το βασικότερο σημείο των συζητήσεων στη Νέα Υόρκη, διότι μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η αντιπροσωπεία μας στη Νέα Υόρκη μπόρεσε να ασχοληθεί με το έγγραφο συμπερασμάτων και τώρα έχουμε και την έκθεση Κάσμαν που χρησιμοποίησε η αντιπροσωπεία μας για να προετοιμάσει τις θέσεις ως προς το τελικό έγγραφο. Το τελικό έγγραφο προωθείται. Πρόκειται για κάπως επώδυνες διαδικασίες, διότι τώρα συζητάμε το έγγραφο. Το έγγραφο από 14 έχει αυξηθεί σε 18 σελίδες, διότι όλες οι αντιπροσωπείες προσέθεσαν ε, σχόλια και όσο περνάει ο χρόνος θα απελτιώνεται. Οι διεκπαιρεωτές μας είπαν ότι θα εισαγάγουν και ορισμένα ε, νέα στοιχεία που δεν αφορούν τους τόχους της χιλιετίας όπως τις κλιματικές αλλαγές έτσι ώστε να διευρύνουμε το πλαίσιο του και να έχουμε μεγαλύτερες ε, επιπτώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι οι διεκπαιρεωτές θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στους στόχους της χιλιετίας. Επίσης θα μιλήσουμε για τον ρόλο των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαμόρφωση των πολιτικών για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, διότι στις ανεπτυγμένες χώρες τα πράγματα δεν έχουν την ίδια εμβέλεια. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ξέρω ότι αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να προωθηθεί το όλο πλαίσιο μέχρι το 2015 για την επίτευξη αυτών των ε, στόχων. Άρα δεν με ενδιαφέρει η έκβαση του εγγράφου. Το έγγραφο θα είναι πολύ καλό και θα αντικατοπτρίζει την έκθεση Κάσμαν και τη θέση της Επιτροπής. Επίσης θα υπάρχει ένας διχασμός βορρά-νότου, διότι δυστυχώς δεν έχουμε ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις για το 2010. Κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε, άρα θα υπάρξουν ε, ορισμένες εντάσεις όμως θα είναι επιτυχής πιστεύω η διάσκεψη κορυφής. Στην Επιτροπή πιστεύω ότι θα έχουμε θετική έκβαση και εργαζόμαστε επί τεσσάρων εγγραφών. Το ένα είναι η πράσινη βίβλος για μια νέα συνένεση για την ανάπτυξη. Να δούμε τι γίνεται μετά το 2005, πώς μπορούμε να αλλάξουμε για μια καλύτερη αναπτυξιακή συνεργασία, τονίζοντας την υγεία, την εκπαίδευση, αλλά όχι όπως κάνουμε συνήθως να μιλήσουμε για την ανάπτυξη, για την εργασία, κατά τρόπο ώστε να μην υποβαθμίσουμε την υποστήριξη. Μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις με την Αφρική και με βάση τη συνολική μας θέση θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην Αφρική. Έχει μεγάλη σημασία πόσο επιτυχής θα σταθούμε στην Αφρική. Επίσης, ε, την πράσινη βίβλο για την δημοσιονομική υποστήριξη είναι ένα έγγραφο που έχει τύχη επικρίσεων και δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία κατά την διαδικασία και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκλίνουμε σε αυτή τη μορφή υποστήριξης. Επίσης, ως προς την δημόσια διαβούλευση για το, τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά και να ακολουθήσουμε το πνεύμα που θα πρέπει να μας διέπει πριν από την διάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο ενωμένη, πιο αποδοτική και θα πρέπει να λογοδοτεί περισσότερο. Και εμείς θα πρέπει να λογοδοτούμε περισσότερο, να είμαστε υπόλογοι έναντι του κόσμου σε σχέση με τις υποσχέσεις μας. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω έχει ως εξής. Προετοιμάζουμε τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής για τα τέλη Νοεμβρίου. Έχουν αποσταλεί οι προσκλήσεις και προετοιμάζουμε και την ημερήσια διάταξη. Πιστεύω ότι θα είναι μια επιτυχής διάσκεψη έτσι ώστε να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση με την Αφρική και να φτάσουμε σε πιο απτά αποτελέσματα. Θα σταματήσω εδώ έτσι ώστε οι βουλευτές να μπορέσουν να γνωμοδοτήσουν και να μου υποβάλουν ερωτήσεις. Γιατί θα ήταν κρίμα να μην έχουμε αρκετό χρόνο για τις ερωταποκρίσεις. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, παρατήρησα ότι δεν είχατε καθόλου σημειώσεις κατά την εισήγησή σας και αυτό δείχνει πόσο ε, ενθαρρυντικά είναι όλα όσα μας είπατε. Ο κύριος Μπέρμαν είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις παρατηρήσεις που μόλις κάνατε. Τρεις, ε, τρία σχόλια θα κάνω σύντομα, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να απαντήσετε αμέσως. Πρώτον, δεν μας μιλήσατε καθόλου για την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ε, ε, δομή της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να, μας, να τοποθετηθείτε για τη θέση που διαπραγματεύτηκε το Κοινοβούλιο σχετικά με τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Εμείς με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίσαμε τη θέση του Κοινοβουλίου ε, και έχετε νέες ευθύνε ε, σε μεγάλο βαθμό χάρη στο Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και θα θέλαμε να τοποθετηθείτε από αυτού. Δεύτερον, για αυτή τη νέα συνένεση για τα αναπτυξιακά ζητήματα θα μπορούσατε να εισέλθετε σε λεπτομέρειες. Ε, σας παρακαλούμε, τι θέλετε να αλλάξετε, τι θέλετε να βελτιώσετε στην φυστάμενη συνένεση ε, νομίζω ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους ε, στα ευπαθή, στις ευπαθείς ε, χώρες. Υπάρχει κάποια νέα στρατηγική και τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Και δεν είμαι ο μόνος στην αίθουσα που έχω συμμετάσχει σε διάφορες αποστολές, παρατηρη... αποστολές παρατηρητών στην Αιθιοπία. και στο Αφγανιστάν ε, έχει, νόημα, έχει νόημα να υπάρχουν τέτοιες αποστολές παρατηρητών εφόσον δεν υπάρχει follow-up, δεν δίνεται κάποια συνέχεια. Πώς μπορεί να το αλλάξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αν δεν υπάρχει υλοποίηση των συστάσεων που επονούμε μετά την, ε, το πέρας των αποστολών, έχει αυτό κάποιο νόημα. Ε, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη, τώρα που καταλήγουμε στη νέα συνένεση. Ε, τώρα, για την αναστολή τη διάθεση κονδυλίων 600 ε, ε, εκατομμυρίων ευρώ για το Αφγανιστάν, μπορείτε να μας δω, αιτιολογήσετε την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ανακοινωθέν τύπου. μιλήσατε για μια στάση αναμονή που τηρείται μέχρι να λάβει αποφάσει η αφγανική κυβέρνηση. Ε, ενώ εσείς έχετε επιμείνει στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ε, η αναστολή έχει κάποια σχέση με την πίεση ενδεχομένως που ασκείται στην αφγανική κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Ε, θα με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος να αιτιολογήσετε αυτή την απόφαση της Επιτροπής. Πρόεδρος, πολύ καλές οι ερωτήσεις σας και σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ε, επανέρχομαι με την ίδια ερώτηση την οποία έκανα και προηγουμένως, δηλαδή πώς ε, τοποθετούμαστε έναντι άλλων χωρών όπως η Κίνα. Ε, δηλαδή υπάρχουν προκλήσεις μήπως συνδυάζουν τη βοήθειά τους με θέματα διαφορετικά και όχι με τα ανθρώπινα δικαιώματα τι γίνεται με τη συνεργασία που υπάρχει επί του θέματος. Ευχαριστώ. Τώρα ζητώ τον κύριο Κάσμαν να σχολιάσει και μετά θα παρακαλέσω τον Επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρουσίαση και τη δήλωση που έκανε, κυρίως η αναφορά που έκανε στο ψήφισμα για τους στόχους της χιλιετίας ε, της περασμένης εβδομάδας στο Στρασβούργο. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε, ε, παρακαλούμε, τις συστάσεις που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγώ θεωρώ ότι ε, αφαιρέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίηση των μέτρων και αυτό το βρίσκω ανησυχητικό. Η Επιτροπή όπως και το Κοινοβούλιο επιθυμεί τα κράτη-μέλη να τηρούν ε, τη δέσμευσή τους ε, για το 1,7% του καθάριστου εγχώριου εισοδήματος. Εάν δεν έχουμε μηχανισμό παρακολούθησης πώς ακριβώς θα κατοχυρώσουμε τη λογοδοσία των κρατών μελών. Για το αιαρινό πακέτο τώρα, ε, και τη θέση του Κοινοβουλίου για τους στόχους της χιλιετίας. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα αποτελεσματικό αμάλγαμα και αποτελεσματική, αποτελεσματικός ε, δρόμος για να προχωρήσουμε. Ε, κοιτάξτε, στις διαπραγματεύσεις θα υπάρξει συμπεφωνημένη θέση που θα πηχεί και τα σημεία της έκθεσής μου και του ερηνού πακέτου. Ε, θα ε, ακουστεί ενιαία φωνή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις ή μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση από πλευράς των κρατών μελών. Μπορεί να εκφράσουν δικές τους θέσεις. Αναφερθήκατε επίσης στη σημασία των κλιματικών αλλαγών και την άμεση συνέπεια που έχουν οι κλιματικές αλλαγές στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για τη μείωση της στόχιας, για την υγεία και για, ε, για τα υγειονομικά συστήματα. όπως θα έλεγε η Βαρόνια στον ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωματών πρέπει να ε, χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις μας. Ε, θα πρέπει να λογοδοτούν οι εταίροι μας και τονίζω τη λέξη εταίροι γιατί είναι ίσοι, ισότιμοι εταίροι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να διαχειρίζονται οι ίδιες ε, τα προγράμματα ε, και θα πρέπει να ε, παίρνουν και οι ίδιες την απόφαση και να χειρίζονται το πρόβλημα. Οπότε αυτό το, θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις δράσεις μας και αυτό πρέπει να αναφέρεται και στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ε, ήμουν επικεφαλής ε, της ομάδας παρατηρητών για τις εκλογές ε, και με αυτή την ιδιότητα θα τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Μπίρμαν ότι δεν είναι ευχάριστο να συμμετάσχει κανείς σε αυτές τις αποστολές και κυρίως να είναι επικεφαλής αποστολής παρατηρητών για τις εκλογές. Ε, όταν εκπονείται έκθεση ένα χρόνο ή 18 μήνες μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και θα πρέπει να είναι χρήσιμη η έκθεση, ούτως ώστε ε, να υπάρχει συνοχή, να δίνεται συνέχεια, ούτω ώστε όταν ε, προκύπτουν εκλογές ε, μετά την έκθεση των παρατηρητών να έχουμε ένα σχέδιο στο οποίο θα αναπέμπουμε, δηλαδή αν εγκρίθηκε από την από την Εκλογική Επιτροπή το σχέδιο που είχαμε αρχικά συμφωνήσει αν ακολουθήθηκε Αυτά και να σας πω ότι έχω και φιάλτες από τότε που πήγα σε αυτές τις αποστολές παρατηρητών. Ξέρετε, εγώ συμμετείχα σε αυτές τις αποστολές γιατί με ενδιαφέρει η έκβαση, αλλά ξέρετε, τελικά διαπιστώνω ότι κάθε άλλο παραέλεγχο έχω επί της έκβασης της αποστολής. Πρόεδρος, ε, έχουμε τρεις ερωτήσεις, ε, μάλλον έχουμε ερωτήσεις από τρεις συναδέλφους, Επίτροπε, για αυτό το πρώτο γύρο. Θέλετε να απαντήσετε. Θα απαντήσω πρώτα στον κύριο Μπίρμαν για την υπηρεσία εξωτερικής δράση. Μα εργαστήκατε με εκπληκτικό τρόπο. Είναι σαφέστατη η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία για την αναπτυξιακή πολιτική. Έχει τουλάχιστον την ίδια βαρύτητα όπως και η διπλωματία στην υπηρεσία εξωτερικής δράση, Οπότε ε, δεν απεισχνάστηκε αν θέλετε ε, αυτή η διάσταση η αναπτυξιακή. Το αντίθετο χρησιμοποιούνται οι συνήθεις διαβλή, αλλά τώρα ε, επιπλέον έχουμε μια συνολική εξωτερική πολιτική ε, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας στη Σομαλία, στο Αφγανιστάν. Οι περιπτώσει που αναφερθήκατε είναι εξαιρέσει, γιατί έχει σημειωθεί πρόοδος για την εξάλληψη τη φτώχεια ε, η διπλωματία και η αναπτυξιακή συνεργασία ε, βαδίζουν εκ παραλίλου και αναμένουμε ε, πολύ θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Τώρα προετοιμάζουμε τα μέτρα σχετικά με το μνημόνιο συμφωνίας και τις διαθεσμικές, τις διοργανικές συμφωνίες οι οποίες θα θέσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλε τι δραστηριότητε. Γιατί ναι, έχω κι εγώ ευθύνε σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερική δράση. Πώ θα επιτελέσουμε τα καθήκοντά μα. Δεν θα. παρέμβουμε αν θέλετε στις ε, δραστηριότητες υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Θα δούμε σε λεπτομέρειες ε, πώς θα γίνει, ε, πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία στο μέλλον. Πάντως η πολιτική συμφωνία είναι ισχυρή και υπάρχει ευρύτατη συνένεση σε όλα τα επίπεδα. Ε, και ε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστώ με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο μέλλον. Ε, τώρα για την αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε την πράσινη βίβλο και το θέμα, όπως είπατε και εσείς σωστά, είναι να δούμε πώς θα υπάρξει ενεργός εμπλοκή για τα αναπτυξιακά ζητήματα πρώτα απ' όλα έχουμε αποδώσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στους στόχους της χιλιετίας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Με Α υποθέσουμε ότι θα εγκριθεί το σχετικό έγγραφο. Ε, δηλαδή, η διεθνή κοινότητα συμφωνεί. Υπάρχουν πολλές χώρες που συμφωνούν ότι πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί για να επιτευχθούν οι στόχοι. Δεν, μπορούν, δεν μπορούμε να αποτύχουμε ε, σε καμία περίπτωση. Κυρίως θα μιλάμε για την μείωση της στόχιας και για οι ευπαθείς χώρας. Μα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το παρελθόν και το αναγνωρίζουμε. Ε, δηλαδή μπορεί να επιτύχετε τους στόχους ε, για τις χώρες μεσαίου εισοδήματο, αλλά για τις φτωχότερε χώρες, ε, για τις ευπαθέστερε χώρες αν δεν επιτύχετε τους στόχους τότε αυτόματα δεν θα επιτύχετε τα επιδιωκόμενα ποσοστά για την μείωση τη φτώχεια. Ε, υπάρχει αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την σημασία των στόχων της χιλιετίας ε, στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, τώρα για τις κλιματικές αλλαγές έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ναι, θα μπορούσαμε να αναλάβουμε μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Καλή είναι η συνένεση, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα ήθελα εγώ θα ήθελα να έχει την ισχύ νόμου, αν θέλετε, η συμφωνία. Δεν θέλουμε ε, μόνο να συζητούμε σε χώρες... Ε, θέλουμε να εφαρμοστεί ε, το κοινοτικό και ε, κεκτημένο να εφαρμοστεί αυτή η συνένεση σε όλες τις χώρες και να έχουμε τα απαιτούμενα μέσα για να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των μέτρων μέσα στη στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας και μέσα στο πνεύμα της διάσκεψης για τους στόχους της χιλιετίας νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την αναδεξιακή πολιτική και να έχουμε μεγαλύτερη λογοδοσία. Ε, ζητώ συγγνώμη Επίτροπε, την πράσινη βίβλο πότε θα την έχουμε. Ε, απάντηση. Ε, στις 13 Οκτωβρίου μάλλον θα εγκριθεί. Αυτό έχει προβλεφθεί και ε, το επιτελείο μου ε, θα ζητήσει να διαβιβαστεί ευθύ αμέσω στο Κοινοβούλιο. Μόλι περατωθεί η διεπηρεσιακή διαβούλευση, το Σεπτέμβρη θα εκδοθεί η πράσινη βίβλος. Θα δούμε τι θα πει η κοινή γνώμη. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε τη διαδικασία μόνο για να την ανοίξουμε. Θα ακούσουμε τι απόψει όλων, το ώστε ε, να βελτιώσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό είναι ο στόχο. 3,9 ε, εκατομμύρια λείπουν από το Αφγανιστάν για να περάσω στο επόμενο θέμα. Συγγνώμη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια κρατιαή βάση στο Αφγανιστάν για να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση. Ε, πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αλλά όχι μόνο. Ξέρετε, όταν διοχετεύουμε εμείς ένα δίσε ε, το χρόνο και τέσσερα δις φεύγουν από τη χώρα, κάτι δεν πάει καλά. Ε, πρέπει να μένουν εκεί τα λεφτά, όχι να φεύγουν από τη χώρα. Γι' αυτό και αναστήλαμε τη χρηματοδότηση προσωρινά, το τονίζω. εθά, ότι δεν είναι υδατοστεγή τα προγράμματά μας και υπάρχει κάποια διαρροή. Μόνο γι' αυτό το λόγο αναστήλαμε τη χρηματοδότηση. Για την Κίνα τώρα. Με τη διάσκεψη για τους στόχους της χιλιετίας μπορεί να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις η Κίνα. Ε, η Κίνα ακολουθεί την ομάδα των 77 χωρών συνήθως, των 77 αναπτυσσόμενων χωρών. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο η Κίνα γιατί από τη μία ακολουθεί την ομάδα των 77, από την άλλη θα αναπτυγμένες χώρες, είναι λίγο ε, αμφίσιμη. Αλλά βέβαια ε, έχουμε και κοινά συμφέροντα με την Κίνα. Συνεργαζόμαστε με την ε, Κίνα και εν γέννη συμφωνούμε ε, για τον προσανατολισμό. Οπότε, αν εγκριθεί το τελικό κείμενο, θα είναι δεσμευτικό και για την Κίνα και για όλους μας. Τώρα φτάνω στα σχόλια του κυρίου Κάσμαν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία πρέπει να χαρακτηρίζουν όλε τι πολιτικέ μα. Είπατε, μα αυτό είναι και το ε, λεπτό σημείο των διαπραγματεύσεων, το δύσκολο σημείο αν, υπάρχουν, αν κατοχυρώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και η δημοκρατία και συμμετέχουν όλοι στην αναπτυξιακή συνεργασία ακολουθώντας τις αρχές της δημοκρατίας μόνο τότε θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και φυσικά θα πρέπει να έχουμε προβλέψει όταν παρεκκλίνουν από αυτήν την οδό κάποιες χώρες. Πιστεύω ότι οι διαπραγματευτές ε, μπορούν ε, να επιτύχουν αυτά που επιδιώκουν για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την έγκριση της έκθεσης Κάσμαν ναι, και από την έγκριση της κοινή θέση, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει διάφορες ε, συνεδριάσεις συντονισμού στη Νέα Υόρκη και ανέκαθεν υπήρχε ομοφωνία. Δηλαδή εκφράζεται με ενιαία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή βάση και Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στι διαπραγματεύσει, αλλά για να, ε, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρετε εσεί στην έκθεσή σα και στην κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και κόκκινε γραμμέ ε, που δεν μπορούμε φυσικά να υπερβούμε και από αυτό το έγγραφο θα προκύψει ένα θεματολόγιο δράση που απηχεί όμω σε μεγάλο βαθμό και τη θέση, την κοινή θέση του Συμβουλίου και την έκθεση του Κοινοβουλίου. Ευελπιστώ ότι θα τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσει για τι αποστολέ παρατηρητών για τι εκλογές. Ε, είναι εξαιρετικά αξιόλογο αυτό που κάνετε γιατί υπηρετείτε τη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα. Αντιλαμβάνομαι πόσο περίπλοκο είναι το έργο σας γιατί τι είναι, σαν να είσαστε διαιτητές στο παγκόσμιο κύπελο. Κανεί δεν σα θέλει, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Ολλονδοί, ούτε οι Οπαδοί. Όλοι μισούν τους διαιτητές. Μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό. Ε, ό,τι και να κάνετε θα σας πούνε δεν το κάνετε αρκετά καλά. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκθέσεις των αποστολών η εκπρόσωπο εκπρόσωπος θα πρέπει, και θα τη το πω, να δώσει μια συνέχεια σε αυτέ τι εκθέσεις. Είναι λογικό εφόσον έχετε μεταβεί στη χώρα, έχετε παρατηρήσει εκλογέ, εκλογές. Ε, πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσεις ε, με τις αποστολής. Ε, για να γνωρίζουμε και πώς ε, έχει η κατάσταση, ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούν. Δεν λέω ότι θα ε, εφαρμοστούν οι συστάσεις 100%. Αλλά μην ξεχνάτε και τις διαπραγματεύσεις του άρθρου 96, όπου προβλέπεται η λογοδοσία και ορισμένες φορές δεν επιτυγχάνουμε τα 100% αλλά το προσεγγίζουμε. Πάντως ε, θα αποταθώ στην ύπατη εκπρόσωπο ούτω ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό στο αίτημα. Νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα, λογική ιδέα γιατί είναι αξιόλογο το έργο των αποστολών των παρατηρητών. Και ε, ξέρετε είναι και συνενετικές οι προτάσεις σας. Ε, δεν είναι ότι το λέει ο Κάσμεν, το λέει ο Είναι συνενετικό η συνενετική θέση που ε, απορρέει από την ε, αποστολή. Δηλαδή προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί η χώρα και άρα θα πρέπει να ε, εξετάζουμε δεόντως τις εκθέσεις αυτές. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ποιος θέλει να ξεκινήσει το δεύτερο γύρο, ο κύριος Γκιόρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία στην αίθουσα του Επιτρόπου Πίμπαλτς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε έναν συνομιλητή ο οποίος μας σέβεται και είναι διαθέσιμος όπως άλλωστε όλοι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι παρίστανται στις συνεδριάσεις. Για να σας πω όμως την αλήθεια, πλέον δεν έχουμε συνομιλητές στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών. Και νομίζω ότι αυτό μας αποδυναμώνει θεσμικά. Και η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη για πολλούς λόγους. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος θεωρεί εδώ ότι μας κοροϊδεύουν, για να σας πω τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πρώτη φορά που δεν μας παρουσιάζουν πλέον τις ε, προτεραιότητες ε, της Προεδρίας στην Επιτροπή μας. Δεν φαίνεται να είναι τελεσίδικα αποφασισμένο το θέμα ε, ή η κυρία Άστον ή η Βελγική Προεδρία θα πρέπει να έρθουν. Θα θέλω όμως να ξέρω αν αυτό το Σαββατό ε, το εξάμεινο θα έχουμε δικαίωμα να ακούσουμε τις θέσεις της Προεδρίας. Δεν είναι δικιά σας δουλειά αυτό. Εσείς μας, λένε, ε, μας λέτε αυτά που έχετε να μας πείτε ε, με την ιδιότητα του Επιτρόπου και είναι πολύ καλά και θα πάμε μακριά μαζί. Αλλά αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδυναμώνεται από την έλλειψη ενός συνομιλητή. Και πιστεύω ότι υπάρχει υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κρύβεται πίσω από όλα αυτά και αν σας το λέγω σε εσά είναι διότι έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε την κυρία Άστον Οπότε ίσως εσείς μπορείτε να είστε ο συνομιλητής αυτής της Επιτροπής και να της πείτε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Ή αυτή η ίδια θα έρθει ή ε, θα αναθέσει σε κάποιον, παραδείγματο χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Βελγική Προεδρία, να έρθει να εκφραστεί εν ονόμα του Συμβουλίου. Είμαστε άλλωστε η μόνη ε, επιτροπή η οποία μπορεί βάσει των συνθήκων να συζητήσει για την αναπτυξιακή συνεργασία και να συμβάλλει σε, μια, σε ένα καλύτερο συντονισμό ε, των πολιτικών σύμφωνα με ε, την ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας διότι τίποτα δεν λέει μέσα στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ότι δεν πρέπει να ληφθούν σοβαρά οι επιθυμίες μας. Θέλω λοιπόν να ξέρω αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι διότι διαφορετικά εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να προτείνουμε κάτι ε, πιο δυναμικό και που θα ξεπεράσει την αίθουσα αυτή και θα ήθελα να έχουμε διευκρινήσει σύντομα. Δεύτερο θέμα. Δεν είμαι αντίθετος στην ε, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία ε, και ε, πιστεύω ότι μπορεί να προβελτιώσει τις συνεργειακές δράσεις αλλά θα ήθελα να τονίσω τις public and private partnerships, διότι δεν τις συζητάμε αρκετά και εγώ τις ανέφερα σήμερα το πρωί, διότι στην Αφρική όταν υπάρχει αύξηση 5% πρέπει ε, να αφαιρέσουμε την ε, πολύ ψηλή θνησιμότητα και άρα ε, ε, ε, αν όλα αυτά γίνουν η ανάπτυξη μηδενίζεται και χρειάζεται να υπάρχει μία ανάπτυξη για να μπορέσει κανείς να κάνει μία ανακατανομή και να αντεπεξέλθει της φτώχειας και όλων των προβλημάτων που έχουν σχέση με τα, τους στόχους της χιλιετηρίδας σχετικά με την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό και μπορείτε να μας πείτε τι αναμένετε από τους υπουργούς των κρατών μελών, από τους υπευθύνους συνεργασίες, πώς η Επιτροπή ε, θέλει να αναπτύξει ή να επιζητήσει συνέργειες με ε, τη ε, Εθνικά Γραφή Ανάπτυξης στα πλαίσια των κοινών προγραμμάτων τα οποία μπορεί να διευρυνθούν στην Επιτροπή εάν ε, συμπληρώνει κανείς περισσότερο τις ιδιότητες των 28 συμμετεχόντων και τέλος όσον αφορά το συντονισμό των πολιτικών γενικώ. Πώς θα τοποθετηθείτε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε και να δούμε πώς θα προωθήσουμε το γεκτημένο του 2005. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να συνδυάσετε αυτή τη συνένεση με την ενίσχυση ε, του θεσμικού πυλώνα για την ανάπτυξη και καταλήγω με αυτά που είπα και στην αρχή, δηλαδή ότι δεν πρέπει να πάψουμε να επαγρυπνούμε μπροστά στον κίνδυνο ο οποίος είναι ουσιαστικός και δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε το μαργαριτάρι των ε, ευρωπαϊκών εξωτερικών σχέσεων. Είμαστε ο πρώτος δανειοδότης, κάνουμε εξαιρετικά πράγματα, είμαστε ανθρωπιστές, ε, προβαίνουμε σε ε, αναπτυξιακή βοήθεια βοήθεια και κρυβόμαστε για να μην υπάρξει συνένεση μεταξύ μας. Με λήψη ενός συνομιλητή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σε ε, την παρουσία του Συμβουλίου κατά τρόπον ώστε να μεταδοθεί και το μήνυμά μας προς τα έξω. Και με αυτό τελειώνω διότι στο πλαίσιο αυτό και λόγω της κρίσεως θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν το 2005 το 0,7% ε, και χάνουμε χρόνο να ψάχνουμε ένα τον άλλον. Οπότε αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα με το να διατυπώσουμε μία θετική προοπτική και να προβάλλουμε προς τα έξω το τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι τόσο σημαντικό ώστε θα, απαντήσω στο... θα παρακαλέσω τον ε, Επίτροπο να απαντήσει αμέσως. Όντως η φύση των εξωτερικών σχέσεων έχει αλλάξει και είναι προφανές ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι ε, πλέον ε, στον ε, εναλλασσόμενο κύκλο των έξι μήνων. Δηλαδή η ύπατη εκπρόσωπος δεν μπόρεσε να έρθει τώρα διότι τώρα εξετάζει την συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής. Το Συμβούλιο αντιπροσωπεύετε Η κυρία Άστον είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα έχετε δηλαδή ένα συνομιλητή όπου συγχρόνως είναι εκπρόσωπος και του Συμβουλίου και ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο συνομιλητής του κυρίου Ντέβε, ε, θα κάνει ό,τι τη ζητήσετε και θα συναντήσετε το Συμβούλιο μέσω αυτής. Αλλά ε, συγχρόνως όπως σας έχω πει είναι και συναδελφός μου. Είναι λοιπόν δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι φοράει δύο καπέλα αλλά θα εκπροσωπήσει εδώ την Προεδρία. Ε, το Βέλγιο δεν μπορούσε ε, να εκπροσωπηθεί εδώ, αλλά είπα την ε, εκπρόσωπος η οποία αποφασίζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου ακόμη και σε θέματα αναπτύξεως καθυστερεί μεν λόγω ανηλυμένων καθηκόντων αλλά θα έρθει και θα σας τα παρουσιάσει όλα αυτά. Όσον όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το πράσινο έγγραφο, όπως σας είπα, το αναφέρει, ε, διότι προωθούμε τις ε, ιδιωτικές πρωτοβουλίες στις υποανάπτυξη χώρες και όπως σας είπα ε, στην χώρα μου αυτό το οποίο κάναμε ήταν να συνδυάσουμε ε, την ιδιωτική ιδιοκτησία με την καλή διακυβέρνηση μέσω ενός σταθερού τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν διότι προωθούν τις συνεργασίες αλλά το, η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι ένα από τα στοιχεία. Επίσης, συνένεση. Δεν είναι η συνένεση το ίδιο με αυτή που υπήρχε το 2005. Νομίζω ότι δεν τονίζουμε ακριβώς το ότι κάνουμε και τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Εγώ ευχαρίστως θα ήθελα μέχρι το τέλος της εντολής να υπάρχει ένα κοινοκτικό και εκτιμένο σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια και θα ήθελα να υπάρχει συνένεση η οποία να βασίζεται στην ε, κοινοτική νομοθεσία. Θα, να είμαστε δηλαδή ακόμη καλύτερα γιατί σήμερα και δεν χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε και πρέπει να στείλουμε αυτό το μήνυμα διότι δεν θέλουμε να ε, ε, ε, περιθεροποιήσουμε τα θέματα αυτά. Θέλουμε να προωθήσουμε και τη Λισαβόνα και την συνεργασία για την ανάπτυξη. Για μένα η συνένεση δεν είναι μόνο συμβολική, αλλά ενισχύει την ΕΟ και στην ανάπτυξη της, στην εξέλιξη της αναπτύξης και εκεί θα ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε γιατί ήρθατε εδώ στη συνεδρίασή μας. Εγώ ε, ήμουν ένας από τους βουλευτές που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στην προηγούμενη συνεδρίαση γιατί είχαμε πολύ λίγο χρόνο και οι πρώτοι παρεμβαίνοντες συνήθως έχουν τέσσερα λεπτά, ο δεύτερος γύρος διαθέτει δύο λεπτά και στο τέλος ε, λέμε στα υπόλοιπα μέλη ότι έχουν 15 δευτερόλεπτα για να προωθήσουν ένα ε, διάλογο με τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Τώρα ευτυχώς έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα εντάχει να υποβάλω τρεις-τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ήδη τέθη, δηλαδή ο βαθμός ικανοποίησης από πλευράς Επιτροπής σε σχέση με την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προωθώντας την αναπτυξιακή αυτή δράση μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Άρα όλοι οι συντονιστές και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων έδρασαν από κοινού για να ενισχύσουν την θέση του Επιτρόπου Ανάπτυξης και της αναπτυξιακής πολιτικής μέσα στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Δεύτερον, θα ήθελα να προωθήσετε αυτό των προμαχών θέσεων που προβάλαμε σε σχέση με ορισμένα αιτήματα για νέα μέσα χρηματοδότησης δηλαδή ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια. Ζούμε μία μορφή συγκαταβατικότητας και στα πλαίσια των G20, καθώς και κατά την Παρασκευή του Κανκούν. Στην αρχή, οι G20 ε, είχαν γνωστοποιήσει την ύπαρξη ενός κοινού προβλήματος και τώρα έχουμε την εντύπωση ότι κάθε μπλοκ, κάθε ήπειρος έχει ξεχωριστά προβλήματα άλλοι ως προς το χρέος, άλλοι ως προς τους αναπτυξιακούς ρυθμούς και δεν υπάρχει αυτή η μεταρρυθμιστική βούληση που προέκυψε μετά από τις πρώτες ε, διασκέψεις των ε, G20 και το γεγονός ότι φορολογούνται οι τραπεζικές συναλλαγές ή ο άνθρακας για νέες αναπτυξιακές πολιτικές εντατικών ρυθμών αυτό απομακρύνεται, απομακρύνεται με συγχωρείτε, στον ορίζοντα. Το ίδιο αφορά και το Κανκούν. Νομίζω ότι όλοι οι παρόντες συμμερίζονται μαζί μου ότι εδώ και ένα χρόνο ήμασταν πιο ανήσυχοι για τα αποτελέσματα της Κοπενχάγης από ό,τι είμαστε τώρα ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα του Κανκούν. Διότι η Κοπενχάγη ήταν μια σχετική αποτυχία από πλευράς ε, αναπτυξιακής ε, συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η προτεραιότητα είναι η Αφρική, σίγουρα. Εκεί συγκεντρώνεται ο αποκλεισμό σε τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά ελλείμματα. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε εφάνταστοι και σε άλλες περιφέρειες του κόσμου ιδιαίτερα ως προς την ε, Λατινική Αμερική. Όλοι έχουν χαμηλά ή μέσα εισοδήματα, αλλά σε αυτές τις χώρες υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα και μεγάλη θύλακες φτώχειας και περιθωριοποίησης σε σχέση με τις ε, μειοψηφίες και τις διάφορες φυλές. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε απλά να θεωρήσουμε δεδομένο ε, γεγονός ότι μέτρο είναι το μέσο εισόδημα τη στιγμή που υπάρχουν θύλακες φτώχειας. Υπάρχει και η συνεργασία νότου-νότου και η δυνατότητα ώστε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής που γνωρίζουν καλύτερη κατάσταση να αποτελέσουν σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνεργασία των πιο φτωχών χωρών. Τέλος, ως προς την ΑΕΤ. γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε γενικά ότι η ΑΕΤ είναι μία δοκιμή για την λειτουργία της κοινοτικής πολιτικής, για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την μετάβαση από την αναπτυξιακή βοήθεια στις αναπτυξιακές πολιτικές. Και νομίζω ότι τα τελευταία δεδομένα που προέρχονται και από τα Ηνωμένα Έθνη δείχνουν ότι καταφέραμε πράγματα αλλά βρισκόμαστε πολύ μακριά ως προς την εκπλήρωση ορισμένων παραμέτρων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μάθει το μάθημα της ΑΙΤΙΣ και να προωθήσει την πολυετή αναπτυξιακή βοήθεια και να προσαρμόσει τις αναπτυξιακές πολιτικές σε αυτόν τον προγραμματισμό που πάει πέραν από την κατεπίγουσα βοήθεια που μπορεί να ανακύψει ή πρέπει να αντιμετωπιστεί ανα πάσα στιγμή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κέλλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ δύο σχόλια και ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με το θέμα της χρηματοδότησης. Νομίζω ότι είναι επίγον το θέμα στην περίπτωση της Γερμανίας. Γνωρίζουμε ότι γίνονται κυβερνητικές περικοπές σε θέματα αντιμετώπισης κλιματικών αλλαγών. Και φαίνεται ότι είναι αποδεκτό πια ότι δεν θα φτάσουμε στο στόχο του 0,7%. Αυτό γίνεται αποδεκτό από την κυβέρνηση. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο επίγον είναι το θέμα. Το δεύτερο αφορά την Ευρωπαϊκή Συνένωση για τους αναπτυξιακούς στόχους. Θα πρέπει το πλαίσιο να είναι πιο δεσμευτικό. Αν αρχίσουμε τη διαδικασία τώρα, τότε δεν θα ε, επιτευχθεί η συνένεση μεταρρύθμισης ή αναθεώρησης μέχρι το 2011. Το 2015 είναι πολύ κοντά, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακού στόχους της χιλιετίας και να λέμε ότι κάτι θα κάνουμε το 2015 και το 2015 να τονίσουμε ότι δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Θα πρέπει τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά τους αναπτυξιακούς στόχους της ε, χιλιετίας. Ως προς τις προτεραιότητες για το τρέχον έτος και τα αμέσως επόμενα, και όπως αναφέρετε και στα έγγραφά σας, πολλά θέματα αναφέρθηκαν, αλλά πού αλλού βλέπετε προτεραιότητες ως προς την μεταρρύθμιση της, ε, της ΚΑΠ, την αλλιευτική πολιτική ή άλλους τομείς. Πού βλέπετε να εγγράφονται προτεραιότητες και να πρέπει να παρέμβετε αναπτυξιακά. Πώς αξιολογείτε τη συνάντηση των G20 στο Τορόντο. Γιατί η έκβαση ήταν πολύ κακή από πλευράς αναπτυξιακών στόχων. Συνήθως έχουμε ωραία λόγια και πολύ καλά αριθμητικά στοιχεία. Αυτή τη φορά δεν είχαμε ούτε καν αυτά. Πώς το αξιολογείτε. Επίσης, μιλήσατε για την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Ποιες είναι οι κατευθυντηρίες γραμμές και προς τα πού θα κινηθούμε στη, προς τη σταθεροποίηση. Προβάλλουμε αναπτυξιακούς στόχους. Και το τελευταίο ερώτημα που μου υποβάλλουν και άλλοι ως προς την ΕΙΕΔ, γιατί δεν, δεν, μπορώ να, δεν μπορώ εγώ να δώσω απάντηση. Είναι το εξής. Επειδή είστε υπεύθυνο. για τα στρατηγικά papers, για τις χώρες ΑΚΕ και τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά παράλληλα τα δύο τρίτα ε, εντάσσονται στην ΕΙΕΔ, πώς θα αναλάβετε αυτή την ευθύνη. Φαίνεται αδιανόητο να ανταποκριθείτε σε περισσότερα καθήκοντα με λιγότερο προσωπικό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η μελλοντική εικόνα. Ίσως κάτι προβλέπετε επ' αυτού. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τέλος η Βερονίκ Ντεκάιζερ για τις τελευταίες ερωτήσεις πριν να απαντήσει ο Επίτροπος που θα έχει πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι όπως και ο Σάγλε νιώθω λίγο απογοητευμένη διότι ε, δεν ήρθε κανένας υπουργός από ε, την Βελγική Προεδρία για να μας ε, παρουσιάσει τις θέσεις και να δώσει εξηγήσει ε, και να δηλώσει ότι παραμένει προτεραιότητα η Αφρικανική Ήπειρος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τη Βελική Προεδρία λοιπόν ε, δεν κατάλαβα γιατί δεν ήρθε κανείς στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, Επίτροπε, ε, μας είπατε αν κατάλαβα καλά ότι δεν μπορούσε κανείς να έρθει διότι αυτό είναι θέμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και ανοίξει το πεδίο αρμοδιοτήτων της Βαρόνης Άστον. Ε, ε, εγώ είμαι μεταξύ αυτών που χάρηκαν για τη συγκρότηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και για το διορισμό της Βαρόνης Άστον, αλλά δεν εννοούσαμε φυσικά ότι θα πρέπει, ε, ότι θα ερχόταν κάποιος να μας πει ότι δεν είναι πλέον ζήτημα της αρμοδιότητάς μας. Είναι κρίμα γιατί ε, ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε είναι ένα κενό ε, πέρα από την επίρρωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. έχει νέες αρμοδιότητες ε, η Βαρόνη Άστον για όλα αυτά τα ζητήματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία, για την εξωτερική δράση, αλλά νομίζω ότι ελοχεύει ένας κίνδυνος, θα δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως και ο Σάγλ. Θα θέλαμε να μάθουμε Ποια νέα όθηση θα δοθεί ε, σε όλους αυτούς τους τομείς όπου χρειάζεται μια νέα όθηση και ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά της ε, εναλλασσόμενης προεδρίας, της Βελικής Προεδρίας. Ο Τις Μπίρμαν ε, σωστά είπε ότι χρειάζεται μία συνέχεια, δηλαδή ανάμεσα στις αποστολές παρατηρητών των εκλογών και των ε, πολιτικών που ακολουθεί στη συνέχεια η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση. Στην έκθεση του κυρίου Σαλαφράνκα και, ε, ε, όπου ήμουν στην στην προηγούμενη θητεία για αυτές τις αποστολές αυτό το ζήτημα της παρακολούθησης είχε κεντρική σημασία. Και ακόμη περιμένουμε απάντηση και συσσωρεύονται οι αποστολές, πολλαπλασιάζονται οι επίμαχες υποθέσεις. Να λοιπόν άλλη μια ζώνη που χρειάζεται δουλειά. Και ζητώ συγγνώμη κύριε Πίμπαλξ γιατί σωστά απαντήσατε αλλά κάνατε αυτό τον παραλληλισμό με τη διαιτησία αλλά δεν συμφωνώ γιατί ο διαιτητής ε, σφυρίζει το τέλος του αγώνα αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πάντοτε ε, αποτελεσματικός. Ε, δηλαδή, ε, εμείς δεν μπορούμε, εμείς δεν είμαστε διαιτητές γιατί δεν σφυρίζουμε το τέλος του αγώνα, δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Αγωνιζόμαστε απλώς. Μιλήσαμε επίσης για την Κίνα και αναφερθήκατε στην απαιτούμενη συνεργασία με την Κίνα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αναπτυξιακή πολιτική της ε, Κίνας. Ε, στο Σουδάν τι είδα, μια υπέροχη φυλακή που είχε φτιάξει η Κίνα για άλλα ωφέλη που ε, θα αποκόμιζε. Αυτό είδα στο Σουδάν. Εμείς επιθυμούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να χαρακτηρίζουν την αναπτυξιακή πολιτική και ρωτώ το εξή ποιες ε, διασυνδέσεις υπάρχουν, ποιες Πώ συνδέεται αυτό το ζήτημα με το διεθνές εμπόριο. Μην μου πείτε ότι συντονίζει και αυτό το θέμα η πατή εκπρόσωπο, γιατί δεν νομίζω να τα καταφέρει όλα να τα χειριστεί ταυτόχρονα. Ε, θα ήθελα να μου πείτε πώ. Πώς ε, συνδέονται αυτά τα ζητήματα και πώς πράξη θα αντιμετωπίζετε τις περιπτώσεις πολυεθνικών στη Βιρμανία, στο Σουδάν, ε, η η επωνομαζόμενη corporate justice, η δικαιοσύνη σε επίπεδο εταιριών. Πώς ε, θα ε, υλοποιηθεί, δηλαδή τι θα το αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων, των πολιεθνικών ή μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι στην πράξη. thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ, κυρία Ντεκάιζερ. Ε, έχετε ε, χρόνο, Επίτροπε, όσο χρειάζεστε. Ε, με την ησυχία σας απαντήστε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Τα είπατε πάρα πολύ ευγενικά. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος τώρα για τις ερωτήσεις του κυρίου Γκερέρο. Πολύ με ευχαρίστησαν οι διαπραγματεύσεις για την υπηρεσία εξωτερικής βοηθείας διότι το Κοινοβούλιο προωθεί την ανάπτυξη και ε, ε, η ανάπτυξη αυτή πλέον δεν ε, θα ακολουθεί την άμυνα ή την εξωτερική, τις εξωτερικές σχέσεις και γι' αυτό θα μπορέσει θεσμικά να εγγυηθεί. Ε, αν ρωτήσετε αντίδραση από έναν πολιτικό σαν εμένα ή την είπα το εκπρόσωπο να εφαρμόσουν αυτά έχουμε δυσκολίες αλλά αυτό που επιτύχατε σήμερα είναι εξαιρετικά. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Έχει γίνει κάποια πρόοδος επί του θέματος διότι αντιλαμβάνομαι ότι πριν τέσσερα χρόνια κανείς δεν μιλούσε για αυτή τη χρηματοδότηση. Τώρα όμως θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Η Επιτροπή έχει ε, κάνει δουλειά του θέματος και Ελπίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν οι πηγές της χρηματοδότηση με την διεύθυνσή τους, είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο όσον αφορά την ε, προτεραιότητα της Αφρικής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και δίκιο έχετε σε αυτό. Ε, βέβαια αυτό το οποίο ε, θεωρώ ότι είναι η πρόκληση και καλύπτει το 50% της ανεπτυξιακής βοήθειάς μας είναι η ε, χώρες μέσου εισοδήματος και ελάχι, το υπόλοιπο μόνο εις ε, τις άλλες χώρες. Ε, θα έπρεπε όμως ε, να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να βρούμε συγκεκριμένες μεθόδους προωθήσεως. Είναι πολύ βασικό η συζήτηση αυτή να γίνει τώρα γιατί η επόμενη δημοσιονομική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη λογική. Και αν θέλουμε να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα χρειαζόμαστε και μια κοινή προσέγγιση για τις χώρες μέσου εισοδήματος του θέματος. Τώρα, ε, όσον αφορά την ΙΤ, ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει καλή δουλειά, αλλά είναι δύσκολη δουλειά η ανάπτυξη και ελπίζουμε ότι αν κάτι δεν γίνει τον επόμενο μήνα θα γίνει σε δύο μήνες και από εκεί αρχίζει ο εκνευρισμός αλλά νομίζω ότι είναι βασικό ότι εφαρμόζουμε προγράμματα ε, βέβαια ε, έχουμε δεσμεύσει όχι ένα υπέρογκο ποσό, 200 εκατομμύρια, αλλά κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν. Και εκεί είναι μία περίοδος που δεν βλέπετε να ε, κτίζονται νέα κτίρια, υπάρχουν ε, δυσκολίες αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις δύσκολες προκλήσεις παρόλο που ε, η πρόοδος μας ε, δεν είναι στο επίπεδο που θα επιθυμούσα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα αυτό της ανάπτυξης. Σχετικά με τα σχόλια της κυρίας Δεκάιζερ, ε, πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι ενοτόμες ε, πηγές χρηματοδοτήσεως και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα. Δεν περιμένουμε πολλά, άρα η συνένεση ε, μας ενισχύει σαν οργάνωση για την την ε, ε, ανάπτυξη. Ε, βεβαίως δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι οι στόχοι θα υλοποιηθούν το 2050 αλλά ούτε ότι μπορεί να γίνουν αύριο. Χρειάζεται να εργαστούμε ήδη σήμερα αν θέλουμε να έχουμε σαν στόχο το 2020 και ε, υπάρχουν ορισμένες ανακοινώσεις ε, αλλά πέραν αυτού ευχαρίσω με το προσωπικό μου να έρθω στην Επιτροπή σας και να εξηγήσω πού βρισκόμαστε. Άλλοι τομείς. Κοινή γεωργική πολιτική είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να μας αποσχολήσει η αλληλεία και επίσης το εμπόριο, διότι το εμπόριο είναι ένα τώρα πολύ σημαντικό θέμα, η μετανάστευση και άλλα. Όλα είναι προτεραιότητες ε, για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία και την πρόθεση της ανάπτυξης. Ε, δεν θα βρείτε παραδείγματο χάρη ε, να απουσιάζει η αλληλεία η οποία είναι σημαντική. Σχετικά με το, το ρόντο, θα περίμενα περισσότερα, ε, δεν κατακρίνω τόσο πολύ, αλλά περίμενα περισσότερα. Και τώρα η γαλλική προεδρία που θα αναλάβει την προεδρία του G20, που είναι μια χώρα η οποία ε, προωθεί τους στόχους ελπίζω ότι θα μπορέσει να συμβάλλει και σε διεθνές επίπεδο και σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό. Οι γενικοί μου διευθυντές μου ζητάνε συνέχεια περισσότερο προσωπικό, αλλά η απάντηση είναι σαφής. Ε, πρέπει να κάνετε τη δουλειά που έχετε με το προσωπικό που υπάρχει διότι κανείς δεν θέλει περισσότερο προσωπικό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς μας τα προγράμματά μας να μπορέσουμε να τα διατυπώσουμε σε μέτρο που να μπορούμε να τα ελέγχουμε και το προσωπικό το οποίο διακινείται ε, νομίζω ότι δεν φεύγουν τα δύο τρίτα, φεύγει το εν τρίτον και διατηρούμε τα δύο τρίτα. Δεν διαφέρει πολύ από αυτά που λέτε, αλλά έχουμε το δυναμικό, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν νομίζω ότι ε, υπάρχει οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει περίκοπες προσωπικού. Ε, πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική ε, και η κυρία Άστον στον καινούριο αυτό λόγο αντιλαμβάνεται το ρόλο του Κοινοβουλίου και θα έρθει εδώ. Τώρα όσον αφορά την Προεδρία του Βελγίου ή μετά του, της Ουγγαρίας ε, η αναπτυξιακή πολιτική είναι λιγότερο ίσως ουσιαστική από ότι ε, το ΕΚΟΦΗΝ αλλά είμαστε δεσμευμένοι και θα σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας. Όσον αφορά την ε, παρακολούθηση ε, νομίζω ότι προσπαθούμε και είσαστε λίγο αυστηροί όσον αφορά την Κίνα και τις πολυεθνικές εταιρείες. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσετε και τι θετικό κάνει η Κίνα ε, διότι ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά αλλά υποθέτω ότι οι Κινέζοι θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν καλύτερα τι κάνουν και δεν έχω κάποιο ε, λόγο να κατακρίνω δημοσίως την Κίνα διότι από πλευράς συνεργασίας οι ίδιοι επενδύουν οπότε ανταποκρίνεται σε μία ανάγκη και πρέπει ε, να ε, να ε, παραδείγματος χάρη να προωθήσουμε τα θέματα της παράνομης υλοτομίας και να μην δεχόμαστε να εισάγουμε προϊόντα παράνομης υλοτομίας για να μπορέσουμε να πιέσουμε ε, τους ε, πολίτες των χωρών αυτών να ενδιαφερθούν περισσότερο για ε, την πολιτική συνεργασία και για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Την επόμενη φορά ίσως θα έχω να σας πω περισσότερα επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε ότι ο Επίτροπος δεν είναι μόνο συνομιλητής αλλά και συνεταίρος στη διαδικασία αυτή και είναι μεγάλη χαρά για μένα να τον βλέπω εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. I now have the great Τώρα έχω το μεγάλο προνόμιο να παραχωρήσω θέση του Πρόεδρου στην ε, κυρία Ανίτσι για να μας παρουσιάσει Σανίτσι, συγγνώμη, για να μας παρουσιάσει το επόμενο σημείο. come coordinare, sì. Grazie, grazie infinite. È la prima volta che mi siedo qua. Σας ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά προεδρεύω. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δούμε πώς θα συντονίσουμε τις ε, προτάσεις μας με βάση ε, ένα ε, σχέδιο της Επιτροπής σε σχέση με το auction floor. Βρισκόμαστε στις πρώτο, στο πρώτο δωδεκάμινο δραστηριοτήτων και πολύ συχνά ήταν δύσκολο να ανταποκριθούμε. Συνάντησα πολλούς ανθρώπους που είχαν πολλές ιδέες και θέλαν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. «Εάν παραμείνετε θα σας τραγουδήσω», λέει η πρόεδρος αρκεί να σιωπήσετε. Γνωρίζω τη σημασία της εργασίας μας, γνωρίζω τον κατεπήγοντα χαρακτήρα των εργασιών μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή μας ή να είναι περισσότερο δίκαιοι. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε να, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτό φαίνεται παράδοξο, αλλά ξέρουμε ότι αυτό ισχύει. Θα πρέπει να βρούμε τους πόρους χρηματοδότησης, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συντονισμός. Ναι, μιλάω πολύ γρήγορα, αλλά είμαι πολύ συγκινημένη, διότι, ε, διότι προεδρεύω πρώτη φορά. Θέλετε να τα πω αγγλικά? Όχι, καλά. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να βρεθεί η χρηματοδότηση και πολλές φορές δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ ε, δωρητών και ενδιάμεσων και γι' αυτό υπάρχει διάχυση πόρων. Γι' αυτό ζήτησα να σας μιλήσω για μία πρωτοβουλία που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και εμείς ως μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης μπορούμε να προωθήσουμε το όλο θέμα. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο μέσα στα πλαίσια των δημοπρασιών διαγωνισμών λαμβάνουμε εκατοντάδες προτάσεων για χρηματοδότηση, ανθρωπιστική βοήθεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα προγράμματα αξιολογούνται από την Επιτροπή, αλλά μόνο ένας περιορισμένος αριθμός την χάνει χρηματοδότησης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ως προς τα τρία τελευταία, τις τρεις τελευταίες προτάσεις, φτάσαμε, ε, είχαμε 758 προτάσεις και μόνο 53 χρηματοδοτήθηκαν, δηλαδή κάτω από το 10%. Θέλω να υπογραμμίσω ότι πέρα από αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν και άλλα έτυχαν θετικής αξιολόγησης. Ήταν κατάλληλα δηλαδή προς χρηματοδότηση, όμως δεν χρηματοδοτήθηκαν διότι δεν υπήρχαν πόροι από την Κομισιόν. Οι ετούντες είναι έμπειροι και το ίδιο αφορά και τους φορείς τους η Κομισιόν χρειάζεται χρόνο, προσωπικό και χρήματα για να αξιολογήσει όλα αυτά τα προγράμματα. Εμείς δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι, διότι κατασπαταλείται αυτή η ποιοτική εργασία. Άρα χάνουμε ευκαιρίες παρέμβασης. Γι' αυτό, μιλώντας με τον δόκτορα Ριντόλφη, που είναι εδώ μαζί μας, ο οποίος ήρθε από την Κίνα, είναι πολύ κουρασμένος, αλλά ήρθε παρόλα αυτά. Είναι υπεύθυνο της μονάδας EuroPaid που ασχολείται με το πρόγραμμα DCI και Food Facility. Όταν μου ε, μίλησε για το auction floor, ε, ήταν έκρινα μια πολύ καλή ευκαιρία. Θέλουμε οι επενδυτές, οι χρηματοδότες και οι άμεσα εμπλικόμενοι φορείς να βρουν τις χρηματοδοτήσεις έτσι ώστε να φέρουν το ποιοτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας έχουν διανύμει και δύο έγγραφα όπου βλέπουμε το βασικό περιεχόμενο των προγραμμάτων Oxenfloor. Το πρώτο, το booklet, αφορά τα πολιτισμικά σχέδια για να έχουμε καλύτερη προσπελασιμότητα στον πολιτισμό στις υποανάπτυξη χώρες. Να προωθήσουμε τις πολιτιστικές βιομηχανίες στις χώρες ΑΚΕ 2008-2008 για έργα στις χώρες ΑΚΕ. Τελειώνω, τελειώνω. Το δεύτερο booklet είναι το Food Facility, facility και Option Floor. Έτσι ώστε να δούμε τα σχέδια, τις προτάσεις διαγωνισμού για το Food Facility για να προβάλλουμε τη διατροφική ασφάλεια στις χώρες του τρίτου κόσμου. Με βάση αυτούς τους δωρητές θέλουμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και το συντονισμό πόρων με βάση την ατζέντα της άκρα. Πάλι μιλάω πολύ γρήγορα. Ε, εντάξει, εντάξει. Τελειώνω, τελειώνω έτσι κι αλλιώς. Εμείς εκλεγήκαμε στο κοινοβούλιο αυτό με βάση την προτίμηση της λαϊκής ψήφου καθώς και ε, ε, εκλεγήκαμε από ενώσεις και βιομηχανίες. Θα πρέπει να προωθήσουμε στις χώρες μας αυτό το πολύ ε, σημαντικό πρόγραμμα, να δούμε ποιοι είναι οι ενδυνάμοι δηλαδή δωρητές να γνωρίζουμε ποια είναι τα καλύτερα αναπτυξιακά σχέδια που κατέρτισαν τα κράτη-μέλη, κατάρτισαν τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να φέρουν το κοινοτικό σήμα. Εγώ ως γυναίκα και ως βουλευτής και μέλος αυτής της Επιτροπής αυτό θα ήθελα να προωθήσω και θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να κάνετε κι εσείς το ίδιο και να συνεισφέρετε στο αίσιο πέρας αυτού του εγχειρήματο. Μίλησα πολύ, αλλά είμαι συγκινημένη και θα δώσω το λόγο στο δόκτωρα Ριντόλφη γιατί είναι αρμόδιος και θα μας εξηγήσει πολύ καλύτερα αυτό το πολύ αξιόλογο πρόγραμμα. Όχι, όχι, μόνο τον τραγουδό θέλω χειροκροτήματα, όχι όταν μιλάω. vero? Adesso fa finta di Καλά, καλά. Πείτε, κάν, κάντε ότι δεν με ακούσατε. Εν περιπτώσει μπορούμε να, οργανώσουμε και μία μικρή συναυλία στο Κοινοβούλιο αν θέλετε με έναν συνάδελφο. Κούφιε! Α, ο συνάδελφος ε, δεν είχε τα ακουστικά και δεν με άκουσε. Άρα πού θα πάει το κοντσερτίνο που θέλω με τον συνάδελφο. Του πάλι Ιταλιάνο, αν ragazzi. Grazie. Α, και εσύ θα μιλήσει Ιταλικά. Μπράβο, μπράβο. Καλό παιδί είσαι και εσύ. Ναι δεν μου τα μετέφρασαν αυτά, αλλά ο Ενρίκε μου είπε τι είπατε και νομίζω ότι τώρα πρέπει να αρχίσουμε τη μικρή μας συναυλία. Ο δόκτωρ Ριντόλφι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τζανίκη για αυτή την πρωτοβουλία που δείχνει ότι έχει ένα όραμα για το μέλλον και θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να προβάλλουν τα θέματα αυτά στην εκλογική τους περιφέρεια και στους συνδέσμους που έχουν με τον ιδιωτικό τομέα, με τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να προβάλλουμε αυτό το πρόγραμμα και να μπορέσει να εκτελεστεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ε, καινοτόμο πρόγραμμα. Ο κύριος Πίμπαλξ σας ε, μίλησε για αυτά τα booklets που έχετε μπροστά σας. Θα ήθελα να τα διατρέξετε. Να δείτε αυτό το δείχνει ο μιλητής που αφορά το Food Facility για τη διατροφική ασφάλεια και αυτό το που βλέπετε που είναι τα πολιτιστικά προγράμματα, το πιο ανοιχτόχρωμο όταν οι ευρωπαϊκές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και τα πανεπιστήμια προβάλλουν προγράμματα μέσω του μηχανισμού εκτέλεσης από τη διαδικασία Call for Proposals κάνουν μία επένδυση. Το ίδιο γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την αξιολόγηση αυτών των προτάσεων με αυστηρό τρόπο ανάλογα με, την, με το, τον ενδυνάμει χαρακτήρα εκτέλεσής τους. Αυτά δεν πρέπει να τα πετάμε στον, στον κάλαθο των αχρήστων επειδή δεν έχουμε πόρους. Θα πρέπει εσείς να διαμεσολαβήσατε έτσι ώστε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προγράμματα έτσι ώστε να επενδύσουν σε μία από τις χώρες αυτές και επίσης και ενώσεις, φορείς που θέλουν να αποφύγουν ένα επιπρόσθετο κόστος να προωθήσουν αυτά τα πρόγραμμα. Και εμείς προσφέρουμε το ποιοτικό κοινοτικό σήμα. Δηλαδή ζητούμε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο να δείτε ποιες είναι οι διασύνδέσεις σας και να χρησιμοποιήσετε την εργασία που έχει ήδη γίνει. Να αξιολογηθούν αυτές οι προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τύχουν χορηγιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και ακόμα και από κυβερνήσεις. Πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία. Πέρυσι αναλάβαμε μια τέτοια πρωτοβουλία στον τομέα του περιβάλλοντος με ένα workshop εδώ και σε αυτό το workshop πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολλοί ε, επιχειρηματικοί σύμβουλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτό το auction floor για αυτές τις δημοπρασίες. Ορισμένα προγράμματα πολίθηκαν μέσα σε εισαγωγικά σε οργανώσεις που τα προτείνουν στη συνέχεια αλλού. Άρα έχει σημασία ο προτείνων, δηλαδή το πανεπιστήμιο, η μη κυβερνητική, κατά την έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, και μέχρι όλη την αλυσίδα, μέχρι δηλαδή την ε, τελική υλοποίηση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την διευκόλυνση, όπως τονίσαμε και στο workshop για τα περιβαλλοντικά. Οργανώσαμε ένα speed dating μεταξύ ε, χορηγών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και δεν θέλαμε να επιλέξουμε πέντε ή έξι σχέδια από αυτό το μικρό βιβλιαράκι, αλλά να εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα και τις μη κυβερνητικέ για να προβάλλουν μια εταιρική σχέση συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό το 0,7% του εθνικού ΑΕΠ θα πρέπει να αφορά και τον ιδιωτικό τομέα και αν για μία επιχείρηση μπορεί αυτό το πρόγραμμα να οδηγήσει στην εισδοχή σε μία αγορά, σε market entry δηλαδή, τότε θα μπορέσουμε να προβάλλουμε και αναπτυξιακούς στόχους με βάση τη Συμβουλή του Κοινοβουλίου. Αυτό ακριβώς αποζητούμε έτσι ώστε να εμπλακούν όλοι οι φορείς. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Τζανίκη για αυτή την πρωτοβουλία και είμαι στη διάθεσή σας. Αυτό που μετράει όμως είναι να διαδώσετε αυτό το βιβλιαράκι στου, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε φορείς, εγώ ξέρω ορισμένους ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούν αναπτυξιακά προγράμματα. Άρα θα μπορούσαμε να προβάλλουμε συμπληρωματικά αυτά τα σχέδια. Είναι projects που συμβαδίζουν με την ατζέντα της άκρα και τη δήλωση των Παρισίων. Δηλαδή συμβαδίζουν με τις πολιτικές που προβάλλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια συνοχής μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δωρητών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε δόκτωρα Ριντόλφη. Είδατε, είδατε σας ε, χειροκρότησαν και ας μην τραγουδήσατε. Λοιπόν, τρεις ομιλητές θα παρεύουν. Καταρχήν ο κύριος Μπέρμαν. Χαίρομαι πάντοτε όταν μου μιλάνε Ιταλικά, γιατί με λένε ονορεύολε και μου αρέσει πάρα πολύ, αξιότιμε δηλαδή κύριε Honorable, πολύ ωραία ακούγεται. Rien Σας ευχαριστούμε για αυτά τα δύο φυλάδια, για αυτά τα δύο εγχειρίδια. Όταν όμως μιλάτε για αυτό το ε, food facility, υπάρχουν 84 προγράμματα που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, 133 που έχουν χρηματοδοτηθεί και πόσα λοιπόν δεν έχουν εγκριθεί, πόσα ε, α, έχουν απορριφθεί μέσω αυτού του διαγωνισμού. Ποιος, ε, με ποιο τρόπο επιλέγησαν τα προγράμματα. Βλέπω πόσο ε, όμορφη, πόσο καλή είναι η διαδικασία, δύσκολο έργο, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες ε, σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. έχει ολοκληρωθεί δε, το food facility. Έχει περατωθεί ή θα δοθεί κάποια συνέχεια. Αυτά θα ήθελα να ξέρω. Diamo, diamo la parola, che sto la parola. Allora non devo dire onorevole ma il signor Cashman κύριος Κάσμαν γίνησε το, ζήτησε το λόγο. Προτιμάτε το ονορεύολο ή το Μίστερ Κάσμαν. Ονορεύολο, ονορεύολο κι εγώ. Ο αξιότιμος φίλος εξ αριστερών ε, θα πρέπει να γνωρίζει ότι όταν ε, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο σε αποκαλεί κάποιος my honorable friend, το αντίθετο εννοεί. Ε, ξέρετε η γλώσσα τελικά, ε, σε όλες τις γλώσσες αυτό που έχει σημασία είναι η χρειά, το χρώμα που αποδίδουμε και πώς χρησιμοποιούμε κάθε λέξη, όχι η ίδια η λέξη. And I think it... Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα προγράμματα και είναι πρότυπη διαδικασία, δηλαδή συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Συζητούμε για κτίρια, για υποδομές. Αυτές οι υποδομές είναι στην καρδιά της ταυτότητάς μας, του πολιτισμού, από μία πλευρά. Και αυτή η πρωτοβουλία για να γίνει το αμάλγαμα ανάμεσα στους ιδιώτες επενδυτές, στους θεσμικούς επενδυτές και άλλους εταίρους στην αναπτυξιακή συνεργασία δείχνει ότι τα προγράμματα θα συνεχιστούν μετά ε, την ε, περαιωσή τους. Μεράτωσή τους, συγγνώμη μετά τον προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας τους θα έχουν και στη συνέχεια επιπτώσεις. Γι' αυτό το Auction Floor, το άλλο πρόγραμμα, εξαιρετική πρωτοβουλία των Δημοπρασιών ε, γιατί ε, ε, εμπλέκονται οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη δική τους ζωή και τη ζωή των άλλων. Μέσω της ιστοσελίδας μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, μέσα επίσης από τις επαφές ε, που έχω, ε, διότι ε, ανήκω στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να προαγάγω το έργο σας. Ε, αυτό το καλό έργο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Ευχαριστούμε που ε, θέσατε υπόψη μας αυτή την καταπληκτική πρωτοβουλία. Γκράτσι Εμίλε. Εγώ σας ε, μίλησα με μεγάλη αγάπη, δηλαδή η εκφορά του λόγου μου αφορούσε ένα βαθύτατο αίσθημα αγάπης, γιατί σας θαυμάζω πραγματικά και σας αγαπώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Άρα... Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι. Άρα ο δόκτωρ Ριντόλφι έχει εκ νέου το λόγο. Thank you, Madam Chairperson. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στα αγγλικά. Αν δεν σας πειράζει για να μιλήσω στον αξιότιμο κύριο Κάσμαν, τον οποίον εκτιμώ. Δηλαδή μπορείτε να αισθάνεστε ότι είσαστε, είσαστε αξιότιμος, honorable μέσω του δημοσιονομικού κανονισμού πρέπει να εφαρμόσουμε διάφανες διαδικασίες επιλογής αλλά υπάρχουν πέραν των προτάσεων πολλές τις οποίες δεν κρατήσαμε ε, διότι θεωρήσαμε ότι δεν ήταν προγράμματα ε, ποιοτικά καλά βέβαια ο ορισμός αυτός είναι σωστός αλλά η διαδικασία διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια και αντιστέκεται εις τις προκλήσεις. Καταρχής σε ένα σημείωμα σε πέντε σελίδες ε, ε, χωρίς να προβεί σε μεγάλη δαπάνη η μη κυβερνητική οργάνωση θέλει, πρέπει να παρουσιάσει τι προσφέρει στο θέμα της επιστημιστικής βοηθείας. Οπότε όταν ε, υπάρχει μία καλή πρόταση και που δεν καλύπτει αυτούς τους τρεις στόχους θεωρήσαμε ότι δεν ήταν επαρκές για να δεκτούμε την πρόταση αυτή και πάμε τώρα στο επόμενο και εδώ ζήτησα από τους συναδέλφους να μου, να βοηθήσουν αλλά ε, από τις 800 προτάσεις τις οποίες ε, λάβαμε κρατήσαμε 250-300 οι οποίες, ε, ε, από τους οποίους ζητήσαμε ε, να προβούν σε πλήρεις δηλώσεις όπου η μη κυβερνητική οργάνωση, το Πανεπιστήμιο θα παρουσιάσει πιο λεπτομερώς τι σκοπεύουν να κάνουν, με ποιους τοπικούς ε, βασικό αξιότιμε κύριε Κάσμαν αν έχετε επιτόπιους συνεργάτες παίρνετε πέντε σημεία παραπάνω αν όχι μηδέν ε, για να υπάρξει δηλαδή συνεργασία επιτόπου. 800 ε, πάνε στις 250, από τις 250 διατηρήσαμε 213, δηλαδή 50-60 ε, τελικώς ε, απερίφθησαν στην τελική φάση. Νομίζω ότι τα κριτήρια έχουν ε, δημοσιευθεί και ήταν σαφή και ε, η κοινότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίοι συμμετείχαν ε, χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα σε πολλά μέρη και πέρυσι το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε. Όσον αφορά το Concord, συζητήσαμε με το Concord την πλατφόρμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα κριτήρια. Και συζητήσαμε και στην Επιτροπή DCI για να μπορέσουμε να αντικατοπτρίσουμε το πνεύμα του κανονισμού σχετικά με την οργάνωση για την ψυχική βοήθεια. Ε, με ρωτάτε, τελείωσε η επιστημιστική βοήθεια. Ε, οργανώθηκε πολύ γρήγορα. Είχε ε, παρουσιαστεί το 2008. Το 2009 εγώ προσωπικά είχα υπογράψει πάνω από 6 εκατομμύρια συμβόλαια, δηλαδή έναν υπέρογκο αριθμό σε ένα χρόνο, μοναδικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, λειτουργήσε αυτή η προσπάθεια να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας, να επιλέξουμε χώρες και ε, να καθορίσουμε τους στόχους στους οποίους θα ε, θέλαμε να συνδράμουμε. Ε, όλες οι δεσμεύσεις και αποφάσεις ελήφθησαν, τώρα γίνονται οι παρουσιάσεις, θα τελειώσουν στο τέλος του επομένου έτους και μετά μέχρι το 2012 θα παρουσιάσουμε την τελική μας έκθεση όπως συμφωνήθηκε στον κανονισμό. Βέβαια έχουμε ήδη ε, δεχθεί τον εσωτερικό έλεγχο και διάφορες εκθέσεις οι οποίες είναι πολύ καλές Βέβαια υπάρχουν προβλήματα, δεν σας το αποκρύπτω, διότι πιέζουμε όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια, διότι το, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι σε μία δόση και προσπαθούμε να έχουμε συνέργειες με τις διεθνείς οργανώσεις για να ξέρουμε πού πάμε. Πλησιάζω προς το τέλος κυρία Πρόεδρε και κύριε Κάσμαν. Έχετε δίκιο. Όντως χαίρομαι για αυτά που είπατε, αυτό ήθελα και εγώ να προωθήσουμε. Δηλαδή γιατί έγινε όλη αυτή η δουλειά, γιατί μία μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε δεν έπρεπε να έχει μία επιπλέον δυνατότητα, μία άλλη ευκαιρία και ε, αν, ε, γιατί δεν μπορούμε να συμβάλλουμε ε, και να δώσουμε την δυνατότητα εις, την, στο Ίδρυμα Rockefeller, Big Gates, δηλαδή θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε και αυτό το συντονισμό. Και όπως είπατε αποδείξαμε ότι υπάρχουν πολλά καλά προγράμματα που προέρχονται από τη βάση ε, της ε, συνεργασίας υπάρχει όντως καλός, ε, καλή συνεργασία και έτσι διαδίδουμε τα καλά νέα και προσπαθούμε να καταρτήσουμε αυτή την αλυσίδα μεταφορά των αξιών που επιζητούμε. Ευχαριστώ. Ας ελπίσουμε να ειδωθούμε στο εγγύς μέλλον και να επιτύχετε. Θα παραμείνετε μαζί σας ή θα φύγετε. Αφού ήρθατε, ναι, ναι, ναι, ήρθατε από την Κίνα πρέπει να πάτε να κοιμηθείτε. Και εμείς δεν έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Τι άλλο έχουμε, τι έχουμε για να βάλω τα γυαλιά μου. Περνάμε στα διάφορα. Υπάρχουν άλλα σημεία προσυζήτηση. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Πρόεδρε, σαν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής θα ήθελα να στείλετε μη ένα επίσημο ο γράμμα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι ε, δυσαρεστηθήκαμε με την απουσία του Συμβουλίου εχθές και ε, σήμερα. Δεν μας άρεσε καθόλου αυτό και προσβλέπουμε στην παρουσία τους στην επόμενη συνεδρίαση. Μιλήσαμε για τον ε, προϋπολογισμό, για τον δημοσιονομικό κανονισμό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως, συναντήσαμε τον Επίτροπο Πίμπαλς. Ε, υπήρχαν διάφορα θέματα όπου θα ήταν απαραίτητη η παρουσία του Συμβουλίου και είναι απαράδεκτο η ε, Προεδρία να δείχνει να διαφορεί τόσο πολύ για το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάνει μια σοβαρή δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Θα ήθελα επίσης να πω και κάτι άλλο που δεν έχει καμία σχέση. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον συνάδελφο Γκερέιρο, διότι τα κατάφερε πολύ καλά η Ιταλία ε, ήταν ε, ε, κτρή, ενώ εσείς όχι. Άρα να συγχαρώ ολόκληρη την Ισπανία, ο κύριος Γκερέιρο. Είμαστε πρωταθλητές για πρώτη φορά, ενώ εσείς το έχετε κερδίσει πολλές φορές και η Ολλανδία το άξιζε δύο από τις τρεις φορές ε, ε, η τέταρτη φορά, εάν ο αντίπαλος δεν είναι η Ισπανία, μπορεί να το κερδίσει. Τη επιτρέπουμε. <laughs> Ναι, πράγματι το αξίζει. Σας ευχαριστώ όλους. Ξέρετε ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 30 Αυγούστου από τις 15 στις 18 και 30. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Γεια σας.